Chers collègues, je vous remercie de prendre place rapidement. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, γιατί κάποιοι συνάδελφοι έχουν και άλλες ψηφοφορίες, όπως ο κύριος Χρυσόγονος, σε άλλες επιτροπές. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε μια αλλαγή της ημερήσιας διάταξης που μας ζήτησαν συνάδελφοι που έχουν άλλες ψηφοφορίες στις 10.30. Ε, συμφωνείτε λοιπόν να αρχίσουμε ήδη με το σημείο 17, δηλαδή κατευθείαν με τις ψηφοφορίες για να μπορέσουν να φύγουν οι συνάδελφοι. Διαφωνείτε? Όχι, ωραία. Αποφασίζουμε λοιπόν, παρακαλώ, τοποθετήστε τις κάρτες σας στη σχισμή και αν δεν έχετε τις κάρτες σας, παρακαλώ να μου το πείτε, να σηκώνετε το χέρι σας ε, για να... Ε, μας δείχνετε την ψήφο σα. και η γραμματεία θα σας λάβει υπόψη. Συμφωνούμε? Δεν είμαστε απολύτω έτοιμοι ακόμη. Παρακαλώ πολύ, καθίστε να αρχίσουμε. Ψηφίζουμε το σημείο 17, έκθεση Σφόμποντα. Έτοιμοι. Τροπολογία 111. Υπέρ. Συγγνώμη, 11 διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λείπουν δύο. Δεν έχετε κάρτα. Ποιος άλλος δεν έχει κάρτα. Πολύ ωραία. Πέρασε. 13 υπέρ. Και ο κύριος Τζαμπάσκι που είναι υπέρ επίσης. 14 υπέρ. 8 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. 12. Υπέρ. Κατά. Ίδιο αποτέλεσμα. 14-8. Είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβω ότι γίνεται. Συγγνώμη, 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Ε, δεν είναι πολύ σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, 13 υπέρ, 8 Κατά. Ευχαριστώ. Και δύο εποχές. Τροπολογία υπαριθμών 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία... Συγγνώμη. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα της ψηφοφορία και τα αποτελέσματα είναι 21 ψήφοι υπέρ, 2 αποχές. Καμία ψήφο κατά. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Έκθεση Σπόμποντα και πάλι. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 15 υπέρ, 8 κατά, καμία αποχή. Λάβαμε υπόψη την ψήφο του κυρίου Τζαμπάσκη. Α, έχετε την κάρτα σα τώρα, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Τροπολογία υπαριθμών 12, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Πολύ ωραία, εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Κανένα πρόβλημα. Τόσο αυθόρμητα το είπατε, δεν μπορώ να σας πω όχι. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Ευχαριστώ πολύ. Αποτελέσματα 12 υπέρ, 11, 11 κατά. Καμία αποχή. Ευχαριστώ πολύ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται. Κανείς δεν θέλει έλεγχο. Εγκρίνεται άρα. Τροπολογία 3. Υπέρ.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 Λοιπόν, ηλεκτρονικώς ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Αποτέλεσμα. 21 ψήφοι υπέρ, 2 αποχές, ε, κανένας ε, δεν ήταν κατά. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην επόμενη μας ψηφοφορία και δίνουμε το λόγο, επειδή μας τον ζήτησε, η κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, απλώς θα ήθελα να παρουσιάσω μια προφορική τροπολογία όχι επί της εκθέσεως γιατί ε, συμφωνήθηκε ε, κατά τον τριμερή τετραμερή διάλογο με το Συμβούλιο και με το ε, δικαστήριο. Απλώς θα ήθελα να πω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη να επιστήσουμε την προσοχή στη σημασία που δίνουμε στο gender mainstreaming. Υπενθυμίζουμε λοιπόν τη σημασία που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ισότητα των φύλων ε, και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου μεταξύ των δικαστών του ε, ε, δικαστηρίου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το επενθυμίζουμε. Θα ήθελα παρόλα αυτά, λέει ο Πρόεδρος, να, να, να το θέσω σε ψηφοφορία υπέρ, κατά, Αποχές; δύο, τρεις αποχές, τρεις αποχές. Και τώρα, Ψηφίζουμε το άρθρο όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη. Πέρας. 16 υπέρ, 4 κατά και 3 αποχές. Επόμενο σημείο Ηλεκτρονικός έλεγχος και το επόμενο. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. 19 υπέρ, δύο κατά, δύο αποχές. Ευχαριστώ. Και τέλος... Το τρίτο κείμενο έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Το 24, α, το 24, μάλιστα. Ψηφίσατε όλοι? Πέρας της ψηφοφορίας. Six 6 υπέρ, 17 κατά. Καμία αποχή. Απορρίπτεται. Oui, vous en prie. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί ψήφισα σε λάθος κείμενο. Έπρεπε να ψηφίσω κατά. Τώρα είναι σαφέ. όμω. τώρα κατάλαβα για ποιο ψηφίζαμε. Ε, εντάξει, θα διορθώσουμε την ψήφο σα. Επόμενη ψηφοφορία αφορά τον προϋπολογισμό. Θα τα ψηφίσουμε όλα μαζί on block. Και καλύτερα να το κάνουμε ηλεκτρονικός για να είμαστε σίγουροι. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 18 υπέρ. 4 κατά και καμία, καμιά αποχή, αν διαβάζω καλά, λέει ο πρόεδρος. Θα δώσω μια στο μηχάνημα μήπως τα γράφει καλύτερα. Πάμε στο 22. Από 32. Amendment. L'amendement numéro. Συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους από την ομάδα των σοσιαλιστών να αποσύρουν την τροπολογία 20 στην οποία ζητούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της για το SUP. για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Εμείς εργαζόμαστε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα επί της συγκεκριμένης ε, νομικής πράξης. Και φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση και θα καταπέσει ούτως ή άλλως η πρόταση. Νομίζω όμως ότι θα ήταν πιο ευγενικό και πιο λογικό να μην μπερδέψουμε τις δύο διαδικασίες. Υπάρχουν πολλές συμβιβαστικέ ε, προτάσεις και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι μια καλή γνωμοδότηση. Δεν θα ήθελα λοιπόν το ΕΛΚ να υποχρεωθεί να καταψηφίσει τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση λόγω της τροπολογίας 20 και μόνο. Μήπως θα μπορούσατε λοιπόν να την αποσύρετε. Τότε θα μπορούσαμε να υπερψηφίσουμε. Κύριε Ρέγνερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς έχουμε πολύ ισχυρή θέση ως ομάδα για το θέμα αυτό, αλλά σε σχέση με τούτη τη γνωμοδότηση ε, μπορούμε να αποσύρουμε την τροπολογία 20. Merci beaucoup. Ε. Ευχαριστώ πολύ για τι αποσαφηνήσεις. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τη συμβιβαστική τροπολογία 3 και μετά να συνεχίσουμε με τον κατάλογο ψηφοφορία. Λοιπόν, 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στη 13. Εμφωνούμε 13. Υπέρ. Κατά. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι, ευχαριστώ πολύ, πέρας. Εντάξει. Α, δεν έχει τελειώσει ψηφοφορία, μα δεν ψηφίσατε όλοι. Τώρα εντάξει. Α, ξανά από την αρχή. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 3 ξανά από την αρχή έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Τώρα τα καταφέραμε όλοι. Κύριε Λεμπρωτό, εντάξει, όλα καλά. Ε, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Πέρασε. Αποτελέσματα. 13 υπέρ, 10 κατά. Καμία, καμία αποχή. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Πάμε στην τροπολογία τη συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστή... Όχι, συγγνώμη. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος της τροπολογίας 15. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 11 υπέρ 12 κατά καμία εποχή απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Α, όχι, όχι. 21. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Έντεκα υπέρ, 12 κατά, καμία αποχή. Τεροπολογία 23 ε, εφόσον η 20 αποσύρθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Αλλά καλύτερα να είμαστε βέβαιοι και να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Πέρας. 12 κατά, 9 υπέρ, καμία αποχή. Απορρίπτεται άρα. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Έναρξη. Πέρασε. 16 υπέρ, 7 κατά. Καμία αποχή εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Και κόντρα. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισε πάντα πέρας. 11 προς 10. Υπέρ. 11 υπέρ 10 κατά, Δύο αποχές. Εγκρίνεται. 37 Δυνατάσεις της χειρός υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Ε, καταπληκτή. Η 39 όμως ψηφίζεται. Η 39 τώρα. 39 υπέρ. Κατά. Μάλλον εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός παρακαλώ. άρχιτε η ψηφοφορία. Πέρας. 18 υπέρ, 5 κατά, 3 αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Δυνατά σε της χειρός υπέρ. Κατά. Υπέρ μάλλον. Κατά δεν είναι σαφέ ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. 19 υπέρ κατά 4 κατά και μια εποχή εγκρίνεται. 58 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Να απαντήσω. Ευχαριστώ. Πέρασε. 12 κατά, 11 υπέρ, 3 αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. ως τις χειρός υπέρ, κατά, αποχές, κρίνεται 4 υπέρ, κατά, δεν κρίνεται Ξέχασα τι αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα τροπολογία. Όχι. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. 19 υπέρ, 4 κατά, 2 κατά και 2 αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Κυρία Ρέντα. Για την επόμενη ε, έκθεση για τα δόμενα πυρία. Ο εισηγητή ε, μου ζήτησε να διαβάσω τη δήλωσή του. Η κυρία Χαουταλά ε, βρίσκεται στην ε, Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη για την ανθρωπιστική κρίση και δεν μπορεί να είναι σήμερα παρούσα, αλλά ευχαριστεί όλου για τι δημιουργικέ και επικοδομητικέ του τροπολογίε, γιατί έτσι τονίζονται, τονίζεται η σημασία αυτή τη διάσκεψη. Υπάρχουν δύο τροπολογίε που έχουν μπει στην έκθεση και έχουν παρουσιαστεί ω προφορικέ τροπολογίε. Η πρώτη, τροπολογία 1, συμπληρώνει την παράγραφο 2 και καλύπτει την τροπολογία 10 του κυρίου Μπούντα, την τροπολογία 11 και την τροπολογία 12 του κυρίου ε, Χρυσόγονου. Ε, η δεύτερη συμβαστική είναι η τροπολογία 2 που συμπληρώνει την παράγραφο 3 και καλύπτει τρεις τροπολογίες, την 18, Κόζα, 19, Μπούντα και 21 του Χρυσόγονου. Ε, αυτές οι δύο τροπολογίες ε, υποστηρίζουν ε, πολύ σημαντικά θέματα τα οποία επίσης μπορεί να τα δεχτεί και η κυρία Χάουταλα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μείνουν έξω σημαντικά πράγματα από την έκθεση. Γι' αυτό έχει πει ότι θα συμπεριληφθούν οι δύο αυτές τροπολογίες στην τελική εκδοχή της έκθεσης και ελπίζει ότι όλοι μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, madame. Nous Σας ευχαριστούμε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 Θα τις το μεταφέρετε, ελπίζω. Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες. Διακόπτουμε για λίγα λεπτά, πέντε λεπτά όχι παραπάνω, για να μπορέσουμε να περάσουμε στις σωστές θέσεις και να συνεχίσουμε με τη συζήτηση. Le sujet suivant portant sur la portabilité. Τα επόμενα θέματα για τη φορητότητα.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 Συνάδελφοι, περιμένοντα ε, να αναλάβει και πάλι ο πρόεδρο τη συνεδρίασή μας, Έρχεται και ο θα μπορέσει να συντονίσει τη συζήτηση. everybody agrees. Yes. Uh, dear colleagues, let us continue. Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε. Ανακοινώνοντας καταρχάς τις αποφάσεις της συνεδρίας των συντονιστών. Καταρχάς, ο κύριος Λεμπρετών αναλαμβάνει εισηγητής για την άρση της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου. Ο κύριος Μαρίνιο Επίντου είναι εισηγητής για την άρση της ασυλίας του κυρίου Γιώργου Γραμματικάκη, ο κύριος Βιέφκα είναι εισηγητής για την ε, υποστήριξη της ε, ασυλίας της Jane Collins. Ο κύριος Καβαντά είναι εισηγητής για την απόσπαση εργαζομένων στα πλαίσια της ε, παροχής υπηρεσιών. Ο κύριος Μαστάλκα αναλαμβάνει εισηγητής για τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας ε, ε, απέναντι στις γυναίκες και την οικιακή βία. Η κυρία Κομοντίνη ε, αναλαμβάνει συγκήτρια για την πολιτιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Χρυσόγονος για την άγρια ζωή και την εμπορία αγριών ζώων. Τώρα η κατανομή των εκκρεμουσών εισηγήσεων και των εισηγητών για το επόμενο εξάμενο έχει ως εξής. Νομική βάση κύριος Καβαντά, επικουρικότητα, κύριος Χρυσόγονος, ε, θέματα αμφισβητούμενα η κυρία Χάουταλα, ε, επιτροπολογία και ε, κατεξότηση πράξη η κυρία Φεράρα και κωδικοποίηση και ρίκα στην αναδιατύπωση η κυρία Μπουτονέ. Επίσης, καταγράφεται ε, η επιθυμία για ψήφισμα για τον κανόνα 153 τον, του ιστορικού κανονισμού για το διηγητικό κόστος για τις επιχειρήσεις για, από τη Σοφή Μοντέλ και τον Φλόριαν Φίλιππο. Αυτά. Και με την έγκρισή σας και τη αιτήση του κυρίου Καρίμ, μήπως μπορούμε τώρα να δούμε το σημείο 7, γιατί ο κύριος Καρίμ έχει κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Οπότε, να δούμε το σημείο 7 και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καρύμ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς και όλους τους συναδέλφους που με διευκολύνετε με αυτόν τον τρόπο, γιατί όντω έχετε δίκιο, υπάρχει ένα χρονικό περιορισμό, έχω λίγο χρονική πίεση. Και πρέπει να ζητήσω και συγγνώμη από του συναδέλφου, γιατί εδώ και κάποιε εβδομάδε ε, ήμουν απόν από το Κοινοβούλιο. Γνωρίζω ότι αρκετοί συνάδελφοι προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή μαζί μου αυτέ τι εβδομάδε. Ελπίζω ότι έχω υπάρξει αρκετό καιρό σε τούτο το κοινοβούλιο ώστε να ξέρω οι συνάδελφοι ότι δεν είναι αυτό ο συνήθι τρόπο με τον οποίο λειτουργώ, αλλά ε, αυτή τη στιγμή αυτό που με κρατάει μακριά είναι το δημοψήφισμα στον Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό ταξίδεψα συγκεκριμένα σήμερα για να κάνω την παρουσίαση σε εσά και θα φύγω πάλι για να επιστρέψω στον Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε σα ευχαριστώ πολύ που με διευκολύνετε και κάνετε, έτσι, δείχνετε την ανοχή σα τι τελευταίε εβδομάδε. Λοιπόν, Έχουμε φτάσει ε, στις 23 Ιουνίου βεβαίως, ε, θα μπορέσω να σας καλέσω όλους για να πω το ελπίζω και ελπίζω να μπορέσω να σας πείσω να με συγχωρέσετε που δεν ήμουν εδώ παρόν για να αντιμετωπίσω τα θέματα όπως ε, έκανα τον προηγούμενο καιρό. Επίσης, να ευχαριστήσω τους αδέλφους που και πάλι μου επέτρεψαν να συνεχίσω ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και από την εθνική αλλά και από την ευρωπαϊκή του πτυχή. Ε, μιλούμε για το θέμα της επικουρικότητας και τη σχετική έκθεση, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Όντως, ε, είναι ένα θέμα πραγματικά πολύ σημαντικό και χαίρομαι που μπορώ να υποβάλω την έκθεση αυτή εκ μέρους της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Για αρκετά χρόνια μελετούμε το θέμα αυτό και πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδες συζητητές μου, γιατί πραγματικά ήταν πολύ επικοδομητική η βάση πάνω στην οποία δουλέψαμε. Υπήρχαν βεβαίω κάποιε διαφωνίε, ε, κάποια διαφορετικά στοιχεία, αλλά ελπίζω ότι όπω θα διαπραγματευτήκαμε στο παρελθόν, θα διαπραγματευτούμε και τώρα όποια διαφορά υπάρχει. Κυρία Ντελβό, ευχαριστώ για τη θέση που πήρατε και επίση να ευχαριστήσω και του ε, συναδέλφου που εδώ και πολλά χρόνια μου δίνουν την στήριξή του έτσι ώστε να μπορέσω να ε, συνεχίσω την δουλειά μου. Την κυρία Νίβλερ, την κυρία Ρέγκλερ, τον κύριο Σβιεύκα τους ευχαριστώ όλους. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα στην έκθεση. Η προηγούμενη έκθεση μου για την επικουρικότητα ε, υπερψηφίστηκε κατά τη διάρκεια της ε, Ολομέλειας του Απριλίου και τώρα θα ήθελα να βασιστώ σε αυτή, ενισχύοντας τις αρχέ της επικουρικότητας και τη αναλογικότητα, ε, αυξάνοντας και τον ρόλο και τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη δική μα την ευρωπαϊκή διαδικασία Λήψη αποφάσεων. Προτείνω λοιπόν τώρα να καθορίσουμε κάποιε από τι ε, προτάσει που θα ήθελα εγώ να συμπεριλάβω στην, στο σχέδιο έκθεση ε, του 2014. Ένα μεγάλο κομμάτι τη προηγούμενη εκθεσή μου ε, αφοσιώνεται κυρίω στην επικουρικότητα και όχι στην αναλογικότητα. Σε τούτη την έκθεση τούτου του έτου θα ήθελα να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην αναλογικότητα μιλώντα βεβαίω και για την επικουρικότητα. Αυτό δηλαδή θα συμπεριλαμβάνει περισσότερου ανάλογου κανόνε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ενισχυμένη αναλογικότητα και για τι ε, αξιολογίε εκτεκτήπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να επικεντρωθούμε στην αξιολόγηση της, ε, του τεστ ε, επικουρικότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι τόσο πολύ στην αναλογικότητα. Η άποψή μου λοιπόν είναι να επικεντρωθούμε κυρίω στο πώ το τεστ αναλογικότητα λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια είναι τα κριτήρια που αξιολογούν αυτές τις προτάσεις. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα θεσμικά όργανα, όπως η Επιτροπή των Περιφερειών, που ελέγχουν τακτικά την επικουρικότητα και τον αντίκτυπο στι περιφερειακέ αρχέ, που είναι επίση σημαντικό όταν μελετούμε θέματα αναλογικότητα τη νομοθεσία για συγκεκριμένου τομεί. Στην έκθεσή μου που υιοθετήθηκε στην ε, Ολομέλεια του Απριλίου υπήρξε μια πρόταση για μια ενδιάμεση αξιολόγηση και ένα ε, έλεγχο επικουρικότητας ε, και έγινε δεκτή. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλή ιδέα να ορίσουμε τώρα ποιο θα είναι το format για αυτό το τεστ επικουρικότητας στην έκθεσή μου. Επίση, θέλω να σα επιβεβαιώσω, συνάδελφοι, ότι εδώ δεν έχω κανένα σκοπό να υπονομεύσω το ρόλο των κρατών μελών να τροποποιούν την νομοθεσία. Αλλά θα πρέπει να, είμαστε, να μπορούμε να ελέγχουμε ότι οι αρχέ τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητας γίνονται σεβαστέ σε όλη τη διάρκεια τη διαδικασία, Γιατί αυτή είναι μια, είναι μια υποχρέωση που απορρέει από τη συνθήκη. Μετά είναι ο ρόλο των... Ε, επαφίεται στους συνομοθέτε για το πώ να προχωρήσουν. Δεδομένης και τη ε, που δίνουν οι εθνικοί ηγέτες στις ε, διαπραγματεύσεις αυτής της ε, νέα συμφωνίας, ε, όπω λέγεται, του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομίζω ότι αυτό βεβαίω ισχύει και για τα 28 κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε όλε αυτέ τι πτυχέ τη επικουρικότητα που καλύπτονται εντό τη έκθεσης. Συναδελφοί, υπάρχει ένα νέο μηχανισμό, ο οποίο δίνει στα Εθνικά Κοινοβούλια τη δυνατότητα να μπλοκάρουν ε, κάποιες προτάσεις της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, αν 16 κρατημέλη αποφασίσουν να συμπράξουν για να τις μπλοκάρουν. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ αυτής της διαδικασίας και χαίρομαι που οι εθνικοί μας ηγέτες κατάφεραν να επιτύχουν και να έχουν την υποστήριξη όλων των κρατών μελών για μια τέτοια σημαντική μεταρρύθμιση. Βεβαίω υπάρχει μια διεύρυνση του, της τρέχουσας ε, περίοδου 8 εβδομάδων σε 12 για την υποβολή αυτής της αίτησης στην οποία επίσης αναφερόμαστε στην προηγούμενη εκθεσή μου ε, και αυτό έγινε γνωστό ως ε, η κόκκινη κάρτα η διαδικασία της κόκκινης κάρτας. Αλλά αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να ε, εμπλέκει τα εθνικά κοινοβούλια στη δική μας την διαδικασία. Και επίσης ε, αποδίδει ένα, μια υποχρέωση στα εθνικά κοινοβούλια να εξασφαλίσουν ότι αξιολογούν αυτό που συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γι' αυτό με, πολλού, πολλούς τρόπους αυτό ε, ουσιαστικά αφαιρεί την ε, δυνατότητα που έχουν να κατηγορούν ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση για μέτρα που δεν έχουν ε, αναλάβει ή ε, είναι πολύ αργά για να τα λάβουν ή που δεν έχουν ασχοληθεί καν για να τα προωθήσουν. Οπότε δίνει ένα, υπάρχει μια ενισχυμένη ευθύνη πλέον στα κράτη-μέλη. Αλλά δεν είναι βέτο, δεν είναι αρνησικηρία. Δεν είχαμε καμία πρόθεση να είναι κάτι τέτοιο, ούτε σε τούτο το κοινοβούλιο, σε όλα τα χρόνια που είμαι εδώ. Δεν είναι βέτο ούτε όπως με τον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβάνονται οι εθνικοί ε, ηγέτες και ούτε εγώ έχω τέτοια πρόθεση. Επίσης, Άλλο ένα ε, σημαντικό μηχανισμό που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα πρέπει να αναθεωρήσει το σύνολο τη Ευρωπαϊκή ε, Νομοθεσία για να συνάδει με την αρχή τη επικουρικότητα και, την... και τη αναλογικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει μια συγκεκριμένη έκθεση που θα συζητηθεί από το Συμβούλιο Υπουργών κάθε χρόνο αν το Συμβούλιο συμφωνήσει ότι η νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα σε εθνικό επίπεδο ή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεπεράσει τα ωριά τη, θα πρέπει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει ή να τροποποιήσει την, ε, την εν λόγω νομοθεσία και επίση η έκθεσή μου τονίζει τη σημασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρέπει πλέον να αντιμετωπίζει τι ανησυχίε των κρατών μελών και μπορεί να συστήσει το πώ τα, Ευρωπα... τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να δράσουν απέναντι σε συγκεκριμένε γνωμοδοτήσει που μπορεί να συζητώνται σε, κάποια, μικρά βήματα, σε, πολύ λίγα κράτη-μέλη. Ε, πρόσφατα συζητήσαμε το θέμα του μηχανισμού της κίτρινης κάρτας για την ε, οδηγία και τις αποσπάσεις. από την ε, εισαγωγή της ε, από το 2009 από τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ξεκινήσει ε, να χρησιμοποιείται ο μηχανισμός αυτός και εγώ αναφέρομαι σε αυτόν στην έκθεσή μου. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση των ανησυχιών των κρατών μελών και αυτό θα πρέπει να το αναλάβει η Κομισιόν. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να ζητήσουμε αν έχουμε συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μας πούν πώς θέλουν να αντιμετωπίσουν, να διαχειριστούν τις ανησυχίες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την οδηγία για τις αποσπάσεις των εργαζομένων. Η επικουρικότητα δεν είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φοβάται είναι σημείο κλειδί ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της και είναι απαραίτητο αν θέλουμε να ε, μειώσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα. Στην, ε, στο τρέχον πολιτικό κλίμα και κυρίως στη δική μου χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, που περιμένει να γίνει το δημοψήφισμα, είναι σημαντικό να δείξουμε στο ευρύ ότι εδώ στις Βρυξέλλες έχουμε την θέληση να ακούσουμε ε, εξασφαλίζοντας ότι θα υπάρξει μετά και νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο εκεί όμως που χρειάζεται. Η επικουρικότητα αυξάνει τον διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια και βεβαίως οδηγεί σε καλύτερη, πιο ε, σωστή νομοθεσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το επικοδομητικό τους πνεύμα και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα που υπέβαλαν οι εν λόγω αρμόδιοι Επιτροπή, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα ε, εκπονούμε νομοθεσία με τον τρόπο με τον οποίο μας περιμένουν και οι πολίτες μας να το κάνουμε. Βεβαίω βεβαίως προσβλέπω στην πρόοδο που θα επιτευχθεί στον φάκελο αυτό και βεβαίως θα επανέλθω σε εσά στο εγγύς μέλλον, ελπίζω έχοντας και το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος μέλος. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θα επανέλθω εδώ, αλλά εν τω μεταξύ η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή για όλους τους συναδέλφους, για να ακούσω τις απόψει τους και όπως και παλαιότερα και τώρα θα προσπαθήσω να καλύψω όσο περισσότερο μπορώ τις απόψει σας και τα θέματα που θέλετε να μου θίξετε στα πλαίσια τη γενικότερη έκθεση μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Να ακούσουμε τώρα τα σχόλια των μελών. questions? Ερωτήματα υπάρχουν. Αν όχι, έχω εγώ ένα σχόλιο. Ένα ερώτημα. Μιλήσατε για τον μηχανισμό της κόκκινης κάρτας και τις 12 εβδομάδες, τη νέα προθεσμία. Κατά την άποψή σας, αυτός ο μηχανισμός της κόκκινης κάρτας περιορίζεται στην αρχή της επικουρικότητας όταν διάβασα εγώ το κείμενο, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι είναι ένας πιο ευρύς μηχανισμός. Δεν ε, στοχεύει μόνο το Συμβούλιο. Νομίζω ότι δεν ε, περιορίζεται μόνο σε ε, αιτιάσεις που έχουν να κάνουν με έλλειψη σεβασμού στην επικουρικότητα. Ε, κύριος Καρύμ, για τους σκοπούς της δικής μου έκθεσης που είναι πολύ συγκεκριμένα στοχευμένη στην επικουρικότητα και την αναλογικότητα, για τους σκοπούς λοιπόν τούτης της έκθεσης, αυτό είναι ο ορισμός εντός του οποίου θα λειτουργήσω εγώ. Ευχαρίστως να δούμε τις ανησυχίες σας αν υπάρχουν από τους συναδέλφους, για πιο ευρύ ε, τομεί, για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να το καλύψουμε αυτό, αλλά δεν θέλω σε καθέ, σε, με κανένα τρόπο να επεκτείνω το, την εντολή που έχω για την ε, έκθεση αυτή ε, σε όρια που δεν θα, που τις επέτρεπα να είναι αποδεκτή πλέον. Ευχαριστώ. Βεβαίω και εγώ προβλέπω στη συνεργασία μας για το θέμα αυτό. Υποστηρίζω και εγώ την ιδέα ότι η επικουρικότητα θα πρέπει να ενισχυθεί, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να είναι λειτουργικό ο μηχανισμό τη κίτρινη κάρτα. Και επίση θεωρώ ότι χρειάζεται αλλαγή στη συνθήκη για να μπορέσει ο μηχανισμό αυτό να λειτουργήσει σωστά. Αλλά ανησυχώ κάπω για αυτή την ε, πολύ ενισχυμένη ατζέντα για την επικουρικότητα, η οποία, την οποία υποστηρίζω, αλλά η οποία μπορεί να, να εμπλέξει ακόμη περισσότερο την εκπόνηση νομοθεσίας. Και αυτή είναι μία από τις ανησυχίες που έχω. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε στο τέλος να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Η κυρία Μπουτονέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Καρύμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις παρατηρήσεις που κατά τη γνώμη μου πηγαίνουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, η έκθεση 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι λίγο επιφανειακή ω συνήθω. Όσον αφορά τι μελέτη, μελέτες αξιολόγηση αντικτύπου, το αποτέλεσμα είναι και πάλι απαράδεκτο. Είναι γεγονό ότι η διατύπωση του πρωτοκόλου 2 είναι πολύ προβληματική, κάτι το οποίο συχνά ε, δημιουργεί μία ε, αιτιολόγηση πάρα πολύ δύσκολη για ε, τα χρήματα που εκταμιεύονται. Πρέπει να γίνονται αξιολόγηση, γίνεται αξιολόγηση αντικτύπου, η οποία ε, πρέπει να είναι σωστή βάσει της επικουρικότητας. Το 50% για το 2012 ε, ε, ανακοινώθηκε για το 2013-2014. Υπάρχει όμως μια διαφορετικά, διαφορά μεταξύ των δύο αριθμών. Είναι σημαντικό ότι αυτές οι αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται ενδιάμεσα, ως ενδιάμεση αναθεώρηση και φυσικά ως προς τα αποτελέσματά τους μπορούν να βελτιωθούν πολύ περισσότερο Όσον αφορά τώρα την αιτιολογημένη γνώμη ε, που πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και στην αρχή της διαδικασίας πρέπει τουλάχιστον να γίνεται ε, σε διάφορες χρονικές στιγμές. Τα κοινοβούλια τα εθνικά πρέπει και εκείνα να συμμετέχουν και να είναι καλύτερα ενημερωμένα επί των διαφόρων διαδικασιών. Το πρόγραμμα της, Κόζας, ε, της ΚΟΖΑΚ 12 με 14 Ιουνίου μόνο ε, δέκα λεπτά θα ε, αφιερώσει σε αυτό το θέμα. Το σύστημα δείχνει σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδιαφέρεται καθόλου για αυτήν την ε, αρχή που θεωρεί ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ε, στοιχείο του δικαίου της. Πρόεδρος, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιαρντίνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όσον αφορά τα εισαγωγικά ε, σχόλια του εισηγητή. Νομίζω ότι ότι το θέμα της αναλογικότητας ε, σωστά τονίζεται. Η επικουρικότητα έχει πολλές φορές εξεταστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Ίσως θα έπρεπε τώρα να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα στην αναλογικότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τμήμα της ε, προσπάθειά τη για καλύτερη νομοθεσία θέλει να εφαρμόσει πλήρω ε, την αρχή τη ε, αναλογικότητα ω τμήμα των μέσων που έχει στη διάθεσή τη για να ρυθμίσει ε, το πόσο. Εντατικέ θα είναι οι προτάσεις που θα κάνει ε, στο άμεσο μέλλον. Είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο του κανονισμού ε, υπάρχουν κάποιες διατάξεις όσον αφορά την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και όσο το, ε, όσο πιο συγκεκριμένοι μπορεί να είμαστε επί αυτών των ζητημάτων, τόσο το καλύτερο. Όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία που ανέφερε κάποιου από του συναδέλφου σα, όσον αφορά την υποβολή του ε, ρυθμιστικού ε, οργάνου που ε, επιβλέπει την ποιότητα των μελετών αξιολόγησης αντικτύπου κατά τη διάρκεια των ετών έχει ενισχυθεί αυτό το συμβούλιο το ρυθμιστικό και κάποιες γενικές διευθύνσεις μπορούν να επανυποβάλουν το σχέδιο μελετών αξιολόγησης αντικτύπου αν θεωρούν ότι η ποιότητα δεν είναι επαρκής. Και ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που, έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που έχετε να αντιμετωπίσετε είναι η έλλειψη της, ε, ε, του σεβασμού της επικουρικότητας. Δεν έχουν από μόνες τους αξία αυτές οι μελέτες, δείχνουν την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και, και του Συμβουλίου του Ρυθμιστικού για, την, για το σεβασμό της επικουρικότητας. Ε, μελετά τη σχέση μεταξύ των μελετών αξιολόγησης ε, μεταξύ δύο ετών για το ίδιο θέμα. Αν υπάρχει μία έλλειψη σεβασμού ε, του, του, της επικουρικότητας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σίγουρα όχι. έχουμε λάβει ε, τα 14 ε, κοινοβούλια έχουν στείλει αιτιολογημένες ε, γνώμες, κάτι το οποίο είναι πάνω από το κατόφλι για να αρχίσει ο μηχανισμός ε, της διαδικασίας ε, της αποκαλούμενης κίτρινης κάρτας και τώρα εμείς αυτό επεξεργαζόμαστε, αυτό ε, συζητούμε. Τρεις τρόποι υπάρχουν βάσει του πρωτοκόλου 2. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει, να διατηρήσει ή να αποσύρει την πρότασή της. Είναι τρίτη φορά στην ιστορία ότι, που υπάρχει τρίτη κάρτα για μία, κίτρινη κάρτα για μία από τις προτάσεις μας. Στις δύο περιπτώσεις μέχρι τώρα η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρώτη φορά απέσυρε την πρότασή της και στη δεύτερη τη διατήρησε Εξηγώντα για ποιο λόγο. Οπότε σε αυτή τη φάση εγώ δεν μπορώ να προβλέψω τι θα αποφασίσει το Σώμα των Επιτρόπων. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όντως έχει κατά κάποιο τρόπο δρομολογηθεί η διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα εξετάζει το περιεχόμενο των ε, Τη αιτιολογημένη γνώμη των 14 ε, κοινοβουλίων. Πρέπει να δούμε ε, το περιεχόμενο λεπτομερώς και στη συνέχεια το Σώμα των Επιτρόπων θα αποφασίσει ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Θέλει ο κύριος Καρίμ να σχολιάσει. Ε, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά. Ε, σε σχέση με αυτά που άκουσα. Ε, δεν μπορώ να συμφωνήσω με όλα όσα άκουσα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ επικοδομητική η πρόθεση, κάτι το οποίο εμένα μου δίνει μια καλή βάση να αρχίσω την εξέταση, τις ευρύτερες ε, ιδέες που τίθενται και να δω τι μπορώ να λάβω υπόψη μου. Πάντως, το... Πάντως ο, ο προορισμός φαίνεται να είναι ο ίδιος σε σχέση με όλα όσα άκουσα από τις διάφορες πολιτικές ομάδες, από την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ε, ελπίζω να τηρήσει την πρόθεση του, την ανακοίνωση που είχε κάνει ο ε, κύριος Τίμερμαν όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του ε, σε σχέση και με το IAA, το οποίο τώρα έχει ξεκινήσει, ελπίζω όχι μόνο να συνεχίσουμε αυτά που έχουμε ήδη επιτύχει, αλλά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και γρήγορα και αποτελεσματικά από το σημείο από όπου βρισκόμαστε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν το ε, σημείο 7 τη ημερήσια διάταξη. Μπορούμε να πάμε στο 15 το οποίο είναι ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τη διασυνοριακή φορητότητα ε, των ε, διαδικτυακών υπηρεσιών περιεχομένου στην εσωτερική αγορά. Κύριε Καβαντά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικές γενικές αρχές που διέπουν το κείμενο. Το σχέδιο γνωμοδότησης, το οποίο ε, σε σύντομα θα σας ε, υποβληθεί, πρέπει να ε, εξυπηρετεί πέντε βασικούς στόχους. Πρώτον, ο κανονισμός της φορητότητας πρέπει να είναι, ε, να ε, ανάλογος με την πραγματικότητα της παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο και επίσης αξιοποίηση του δυναμικού αυτού διασυνοριακά που είναι 29 δισεκατομμύρια μεγάλο ποσοστό ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή η φορητότητα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργεί πρόβλημα στο επίπεδο προστασίας ε, των δικαιωμάτων του δημιουργού και ε, αυτό για το βασικό λόγο γιατί αυτός είναι, αυτή είναι η πηγή της πολιτιστικής δραστηριότητας και του πλούτου και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση αυτός ο πλούτος να περάσει σε άλλα χέρια. Τρίτη αρχή ότι ο σεβασμός της εδαφικότητας ε, πρέπει να ε, καθιερωθεί. Η, φορ, η φορητότητα διασυνοριακή δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει σύγχυση ε, της πρόσβασης στο διαδίκτυο ως προς αυτό. Υπάρχει επίσης ε, η νομική διάσταση που πρέπει να θεωρείται μία εξαίρεση υπέρ της φορητότητας και όχι ένας νέος κανόνας για την τροποποίηση ή τη δημιουργία σύγχυσης σε σχέση με, τη δημιουργία, με την, τα δικαιώματα του δημιουργού. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι υπηρεσιών ε, δεν ε, ε, πρέπει να δουν τα δικαιώματά τους να, ε, θύνουν, να θίγονται και πρέπει η ευελιξία να αυξηθεί. Όσον αφορά τώρα το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, πρέπει να ισχύει αυτόματα όσον αφορά τις υπηρεσίες παροχής περιεχομένου στο διαδίκτυο με πληρωμή γιατί μπορούν να ε, ε, ελέγξουν ε, το κράτος διαμονής των πελατών τους. Συνεπώς, Όσον αφορά τουλάχιστον τις δωρεάν παροχές, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα opt-in, αν οι πάροχοι υπηρεσιών, τέτοιου είδους υπηρεσιών έχουν τα τεχνικά και οικονομικά μέσα για να ε, συμμορφωθούν με τις απαιτήσει του κανονισμού, μπορούν να, να επιλέξουν να ισχύσει ο κανονισμός και για εκείνους. Οι δωρεάν υπηρεσίες πρέπει να έχουν την ελευθερία ε, να διαλέξουν κατά πόσο ε, η φορητότητα της εξυπηρετεί σε σχέση με το μέγεθος του μεριδίου αγοράς τους. Επίσης, και πάλι στο ίδιο θέμα της εφαρμογής, η φορητότητα δεν πρέπει να ε, δημιουργεί κόστος ε, τεράστιου, δυσανάλογο. Η φορητότητα αποτελεί ε, πράγματι κάτι πολύ ε, σημαντικό για πολλούς καταναλωτές ε, και για πολλούς παρόχους στο διαδίκτυο, αλλά δεν πρέπει να αποτελέσει ιδιαίτερο άχθος για τους μικρότερους παίκτες, οι οποίοι είναι και πολλοί στην Ευρώπη και οι δημόσιες υπηρεσίες που θα έχουν πολύ περισσότερες δυσκολίες από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Κάτι ακόμη. Οι ορισμοί το σχέδιο κανονισμού ε, βασίζεται σε δύο βασικές αρχές, τις οποίες πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένα. Το κράτος μέλος διαμονής και η προσωρινή διαμονή σε ένα κράτος μέλος που είναι διαφορετική από τη συνήθη διαμονή ε, για το κράτος μέλος διαμονής. Εγώ καταλαβαίνω ότι μιλάμε για το κράτος μέλος το οποίο ε, ο συνδρομητής έχει τη βασική του ε, διαμονή και ε, στον οποίο, στο οποίο κάνει την κατανάλωση, εκεί διαμένει βασικά. Όσον αφορά την προσωρινή, μία συγκεκριμένη οριοθετημένη διαμονή σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, όχι ε, αόριστη που έχει, κατά την οποία έχει φύγει για προσωπικού ή επαγγελματικούς λόγους από το κράτος μέλος τη συνήθου διαμονής. Μπορεί επίσης να πρόκειται για μία μόνιμη περίοδο ε, για, τη, για, επαγγελματικούς λόγους, αλλά πρέπει να είναι οριοθετημένη και ε, που θα ορίζει μία περίοδο επιστροφής στο κράτο μέλο. Μπορούμε να σκεφτούμε για παράδειγμα του φοιτητέ Εράσμους, για παράδειγμα τους αποσπασμένους. Ε, εν πάση περιπτώσει, καλύπτει σχεδόν όλο τον κόσμο αυτός ο ορισμός. Επίσης, αποκλείεται να να, να υπάρξει ένα όριο χρόνου ε, με αριθμό ε, ημερών, εβδομάδων ή μηνών στον κανονισμό, αν τα κριτήρια ε, επιβεβαίωσης της συνήθους διαμονής είναι αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου ορισμού που ελέγχεται και οριοθετείται αυστηρά. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να υπάρχει ένα όριο για τον καταναλωτή, γιατί μου φαίνεται εντελώς, δεν μου φαίνεται καθόλου ρεαλιστικό ε, και είναι και πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Τρίτη αρχή ε, για την οποία θα ήθελα να αναφέρω κάποιες λεπτομέρειες είναι τα κριτήρια επιβεβαίωσης ε, του κράτους μέλους διαμονής. Τα κριτήρια αυτά για το συνδρομητή πρέπει να συμπεριληφθούν σε έναν κατάλογο ε, που ε, συμπεριλαμβάνει αυστηρά κριτήρια που οι πάροχοι πρέπει να επιλέξουν ε, βάσει του επιχειρηματικού τους και εμπορικού τους μοντέλου από τη μία και ένα άνοιγμα σε κάθε κριτήριο που είναι αντικείμενο προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ του παρόχου και του δικαιούχου που θα έχει ε, τις ίδιες, τα ίδια ηχέγγυα ασφαλείας με τα υπόλοιπα κριτήρια στον κατάλογο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει μία ασφάλεια επαρκής για τους δικαιούχους, χωρίς αυτό βέβαια να ε, μην έχει ο, παροχής, ο παροχέας το δικαίωμα επιλογής του κριτηρίου που είναι ε, το καλύτερο για ε, την αγορά του. Επίσης πρέπει να μπορούμε να προσαρμόζουμε τον κατάλογο με διάφορες, σε διάφορες, για διάφορες καινοτομίες βάσει βέβαια το, της τεχνολογικής εξέλιξης. Συγγνώμη που μακρηγορώ τόσο πολύ. Ο, για το τελευταίο ε, σημείο τώρα που θα ήθελα να ε, θέσω, αυτή τη στιγμή έχει γίνει επιβεβαίωση του κράτους μέλους ε, διαμονής του συνδρομητή τη στιγμή της συνδρομής, τότε ο πάροχος μπορεί να κάνει έναν έλεγχο της διεύθυνσης IP του συνδρομητή για να δει πόσο συχνά χρησιμοποιείται το περιεχόμενο στο διαδίκτυο σε κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους όπου διαμένει κανονικά. Πρόσοχη. Δεν θέλουμε να ε, παρακολουθούμε που πηγαίνει ο καταναλωτής, δεν θέλουμε να κάνουμε γεωγραφικό εντοπισμό συγκεκριμένο, αλλά θέλουμε απλώς να επισημένονται ή να, να, να, επισημαίνεται η χρήση του περιεχομένου εκτός του κράτους μέλους συνήθους διαμονής για να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες και πρέπει να ε, σας υπενθυμίσω ότι ούτως ή άλλως αυτά τα κριτήρια επιβεβαίωσης ε, υπόκεινται ε, στις διατάξεις που έχουν να κάνουν με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, έχουμε ένα πλαίσιο εδώ που μπορεί να λειτουργήσει αρκετά ασφαλώς. Επόμενο σημείο που έχει να κάνει με την εφαρμογή του κανονισμού. Για το σημείο αυτό, αναδρομική ισχύς προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συμβάσεις που έχουν συναυθεί πριν από την εφαρμογή του κανονισμού μου φαίνεται ότι είναι η σωστή κατεύθυνση. Αντιθέτως, παρά το γεγονός ότι προτείνεται μία μεταβατική περίοδος ε, έξι μηνών μέχρι την αρχή της μεταγραφής. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να δώσουμε ένα χρόνο περιθώριο για να γίνει, μπορούν όλοι να προσαρμοστούν. Όσον αφορά τώρα την επιβεβαίωση, τη συγκεκριμένη επιβεβαίωση ε, της φορητότητας, μπορεί να πάρει αυτό πάνω από έξι μήνες, όπως και η ε, συμμόρφωση των συμβάσεων που έχουν συναυθεί πριν από τον κανονισμό, γιατί είναι αρκετά περίπλοκη η οργάνωση που πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο λαμβανωμένης υπόψη της τεχνολογικής προόδου και των απατών που μπορεί να γίνουν. Ε, δεν πρέπει λοιπόν να, υπάρχει, να δημιουργείται πρόβλημα στα συμβαλόμενα μέρη λόγω της εφαρμογής του κανονισμού. Όσον αφορά τώρα ε, το χρονοδιάγραμμα, έχω να σας πω τα εξής τέσσερα πράγματα. Θα ζητηθεί μετάφραση από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 21 Ιουνίου του 2016. Παρακαλώ σημειώστε. 21 Ιουνίου λοιπόν θα ζητήσουμε τη μετάφραση ε, της ε, γνωμοδότησης. Θα συζητήσουμε το περιεχόμενο στις 11 Ιουλίου. Προθεσμία υποβολής τροπολογίων 15 Σεπτεμβρίου και το σχέδιο γνωμοδότησης θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Γιούρη αν όλα πάνε καλά στις 13 ε, Οκτωβρίου. Να σας τα ξαναπώ. Αν θέλετε θα απαντήσω και σε ερωτήσεις βεβαίως αν κάτι δεν καταλάβατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που χρειάστηκε να ε, έχω την προσοχή σας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή που ε, μας ε, έδωσε και το χρονοδιάγραμμα. Εμείς συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα με την πρόταση αυτή. Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κατέστησε σαφές ότι ε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αντιμετώπισης του γεωγραφικού αποκλεισμού του περιεχομένου. Πρέπει να φτάσουμε σε μια σε μια συμφωνία γρήγορα και πολλές από τις γενικές αρχές ε, που ανέφερε ο κύριος Καβαντά μας βρίσκουν σύμφωνους, για παράδειγμα όχι εισαγωγή συγκεκριμένου χρονικού ορίου, για παράδειγμα για τους φοιτητές Εράσμους είναι μία από τις ομάδες που θα μπορούσαν να είναι η βασική δικαιούχοι αυτής της πρότασης, όμως, ε, λόγω των συμφερόντων αυτής της ομάδας, είναι σημαντικό να αποσαφηνίζεται στην πρόταση ότι κάθε πάροχος ε, υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωμένος Για παράδειγμα, αν ένας φοιτητής πηγαίνει από τη Γαλλία στην Ιταλία στο, πρόγραμμα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους δεν είναι ανάγκη να έχει μόνο στη γαλλική αγορά πρόσβαση, αλλά μπορεί να έχει και στην ιταλική αγορά για να μπορεί πούμε να μάθει ε, τη γλώσσα ή να έρθει σε επαφή με την τοπική κουλτούρα. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που βρίσκει σύμφωνη και την Επιτροπή, απλώς πρέπει ίσως με μια αιτιολογική ε, αναφορά να το διευκρινίσουμε. Όσον αφορά τον έλεγχο της διεύθυνσης IP με σκοπό τον έλεγχο του τόπου διανονής. Εκεί δεν συμφωνώ πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι τα κριτήρια τα ίδια της διεύθυνσης IP να είναι ένας τρόπος μέτρησης ε, ή τέλος πάντων επιβεβαίωσης του πού βρίσκεται κάποιος και παράλληλα και επιβεβαίωσης της διαμονής. Γιατί η πρόταση αφορά περιπτώσεις ε, όπου ο τόπος κανονικής διαμονής και συγκεκριμένης διαμονής ε, δεν είναι ο ίδιος. Οπότε δεν συμφωνώ με τη χρήση της διεύθυνσης IP κατά αυτόν τον τρόπο. Επίσης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τακτική επιστροφή στον τόπο διαμονής είναι ένα στοιχείο του τι σημαίνει διαμονή, αλλά το να ελέγχουμε μέσω της διεύθυνσης IP κάτι τέτοιο σημαίνει ότι οι καταναλωτές πρέπει να χρησιμοποιούν την υπηρεσία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διέπονται από τον ε, κανονισμό αυτό. Νομίζω ότι πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την προστασία δεδομένων προκειμένου η έλεγχοι για τους παρόχους να είναι ανάλογοι και να μην δημιουργούν πρόβλημα στην κινητικότητα του χρήστη. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, η διεύθυνση IP είναι επαρκής προκειμένου ο πάροχος υπηρεσίας να δώσει πρόσβαση σε ένα χρήστη όταν ε, ε, βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, οπότε να μην μπερδεύουμε αυτές τις δύο αρχές και να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP ως κριτήριο επιβεβαίωσης του τόπου διαμονής. Υπάρχουν, ε, υπάρχουν και τραπεζικοί λογαριασμοί, η επιστοτική κάρτα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κριτήρια. Πολύ ευκολότερο είναι σήμερα να αλλάξει κανεί τη διεύθυνση IP από το να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό σε μια άλλη χώρα. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν ένα ασφαλέστερος τρόπο να κάνουμε αυτό που θέλουμε και να αποφύγουμε ότι την πρόταση τη δική σας ε, για τη χρήση της διεύθυνσης IP. Συμφωνούμε απολύτως με την αναδρομική ισχύ της πρότασης και ότι οι συμβάσεις δεν ε, πρέπει να συναυθούν εκ νέου. Πιστεύουμε ότι έξι μήνες είναι αρκετά, αρκετοί όμως. Ε, αν δεν υπάρχει λόγος να συναυθεί εκ νέου η σύμβαση, τότε νομίζω ότι η εφαρμογή του κανονισμού για τη συγκεκριμένη σύμβαση θα πρέπει να μπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα. Και αυτό είναι και προς ε, συμφέρον των καταναλωτών. Ε, θα περιμένουμε το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή για να πούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο κύριος Βος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της συναδέλφου Αγγέλη Κανίμπλερ, η οποία δεν μπορεί να είναι σήμερα παρούσα γιατί έχει κάποιες άλλες υποχρεώσεις, οπότε θα ήθελα να διαβάσω κάτι εκ μέρους της και εξ ονόματος λοιπόν της ε, Αγγέλικα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια και, τον, ε, και τους συναδέλφους για τις πολύ καλές προτάσεις τους, για την πρόταση τώρα της φορητότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το online περιεχόμενο. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή. Ουσιαστικά ζούμε σε, έναν, ζούμε σε καιρούς που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό για πολλούς πολίτες και για πολύ σύντομα αλλά και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα να μένουν σε άλλες χώρες και με βάση αυτό λοιπόν δεν μπορούν να απέχουν από, τις, από τα προνόμια που έχουν εντός της χώρας του, Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το θέμα των συνδρομών. Τώρα, κάποιες, ε, κάποια στοιχεία της συναδέλφου Αγγέλη Κανίμπλερ για την πρόταση κανονισμού. Το πρώτο, κατά την άποψή τη, είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι στον κανονισμό, στην πρόταση κανονισμού, μιλούμε για θέματα διασυνοριακής φορητότητας αλλά όχι για θέματα διασυνοριακής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο. Οπότε θα πρέπει να δούμε και το θέμα αυτό. για τις υπηρεσίες ας πούμε, που έχουν ε, γίνει στην ε, Γερμανία, το Sky Sport ας πούμε. Ε, εγώ θα μπορώ, θέλω να μπορώ από την Ισπανία για παράδειγμα να έχω πρόσβαση στο, στις υπηρεσίες αυτές. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να ε, μεταφερθεί και σε άλλους ε, τομείς. Επίσης, ένα δεύτερο σημείο που είναι πολύ σημαντικό είναι ποιο είναι ο ορισμός, αναφέρθηκε βέβαια ήδη, ο ορισμός της, ε, του κράτους μέλους διαμονής. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να τον ορίσουμε πολύ συγκεκριμένα, τον όρο αυτό, και εξετάζουμε ακριβώς αυτό το κράτος μέλος διαμονής είναι ύψιστη προτεραιότητα να έχουμε επίσης μη γραφειοκρατικές διαδικασίες και να έχουμε έναν στέρεο ορισμό και σωστή εξέταση και διερεύνηση του τι σημαίνει κράτος μέλος διαμονής. Τρίτο σημείο, δεν πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο αυτές οι δωρεάν υπηρεσίες, τα free services, να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογή οδηγίας. Στις περισσότερες ε, περιπτώσεις δεν υπάρχουν ε, ε, συμβατικές υποχρεώσεις ε, εξ αυτών που να, να, που μπορούν να επιβεβαιωθούν ή να επαληθευτούν από το κράτος μέλος διαμονής του χρήστη. Και υπάρχει και αυτό το opt-in που θα μπορούσε ίσως να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτές τις δωρεάν υπηρεσίες, τα free services βεβαίως. Προσβλέπουμε με μεγάλη υπομονησία στην συζήτηση που θα γίνει σχετικά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Κιώστερ. Κύριε, ο ο κύριος Κιώστερ. Ναι, ευχαριστώ. Ε, και εμείς χαιρετίζουμε την πρόταση της Κομισιόν για τη φορητότητα του ψηφιακού περιεχομένου και των υπηρεσιών. Είναι πραγματικά σωστή η προσέγγιση έτσι ώστε οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να χρησιμοποιούν διασυνοριακά τι ε, ψηφιακέ υπηρεσίε. Ένα σημείο κλειδί στην πρόταση τη Κομισιόν ε, έγκυται στην στην εσωτερική, στις εσωτερικές υποχρεώσεις που έχουν ε, τις χώρες, δηλαδή τις χώρες στην οποία ζουν οι χρήστες, οι συνδρομητές και αυτό σημαίνει ότι το ε, περιεχόμενο αυτό θα πρέπει να ε, να μπορεί να είναι προσβάσιμο και να υπόκειται στις ίδιες ε, ε, απαιτήσει διασυνοριακά όπως και εντός της χώρας. Χωρίς δηλαδή ο χρήστης να πρέπει να αποκτήσει νέα συνδρομή στην καινούργια χώρα στην οποία, στην οποία ζει. Δεν θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν κανένα είδου περιορισμός, κάτι που μπορεί να γίνει μέσω του σωστού ορισμού του κράτους μέλους διαμονής. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Υποστηρίζω τον ορισμό του κράτους μέλους διαμονής. Μιλούμε για ένα κράτος μέλος όπου ο συνδρομητής ζει, έχει τη συνήθεια διαμονή του και στο οποίο επιστρέφει συχνά. Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να επαληθεύουν, να μπορούν να επαληθεύουν και πρέπει να μπορούν να επαληθεύουν την ε, ε, έδρα του ε, συνδρομητού. Θα πρέπει βεβαίως να είναι ανάλογη ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό και να μην, ξεπερνά, και να μην ξεπερνούν η διασυνοριακή πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο τις απαιτήσει της εγχώριας πρόσβασης. Βεβαίως θα πρέπει πάντα να υπάρχει νομική ασφάλεια, ε, έτσι ώστε να υπάρξει και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ο στόχος του κανονισμού δεν έγκυται στο να ε, πληγούν οι υπάρχουσες ε, άδειε. Αυτό είναι σημαντικό σημείο και για την χρηματοδότηση, για την παραγωγή και για τη διανομή το, της ευρωπαϊκής πολιτιστικής παραγωγής. Άλλο ένα ερώτημα τίθεται σε σχέση με τους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι δεν ζητούν ε, χρήματα για την παροχή υπηρεσιών και αυτοί θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κανονισμό εφόσον εξετάζουν την, ε, το κράτος διαμονής όπως το εξετάζουν και οι πάροχοι υπηρεσιών που ζητούν ε, συνδρομή. Θα πρέπει λοιπόν για όλους τους συμμετέχοντες ο κανονισμός αυτός να έχει ε, λειτουργικές διατάξεις έτσι ώστε όλο και περισσότεροι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να υποφεληθούν από τον κανονισμό αυτό με βάση και τα όσα πρότεινε ο κύριος Καβαντά. Και βεβαίω σε σχέση με τα όσα είπαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι, νομίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή λύση για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μπορούσαμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σμίμαν εκ μέρους της Ολλανδικής Προεδρίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση για τον κανονισμό περιφορητότητα είναι ένα σημαντικό πρωτοβήμα για τη θέσπιση ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Η σήμανση είναι μια από τι πρώτε προτεραιότητε. Η πρόθεση μάλλον τη ενιαία ψηφιακή αγορά είναι από τι πρώτε προτεραιότητε τη Ολλανδική Προεδρία. Και τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα συμφώνησαν με τι προτεραιότητέ μα. Οι εμπειρογνώμονε έχουν εργαστεί εντατικά έκτοτε με προτάσει που συμπεριλαμβάνουν συμβιβαστικά κείμενα. Λόγω χάρη, ε, θέματα που έχουν ήδη εξεταστεί πέντε φορέ στην ε, αρμόδια ομάδα εργασία στο Συμβούλιο και τι αποφάσει που ελήφθησαν στι 26 Απριλίου εκεί. Ε, χάρη στο επικοδομητικό πνεύμα των αντιπροσώπων μεταξύ του, είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε πολύ λίγο χρόνο. Στι 13 Μαου εξευρέθη στο Κοραπέρε συμβαστική λύση και το ερχόμενο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, περιμένουμε να επιβεβαιώσει αυτή τη συμβαστική λύση για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα. Merci, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω απλώς τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους και να σας πω με τρόπο ξεκάθαρο ότι εφόσον πληρωθούν οι συνθήκε που μόλι ανέφερε και το Συμβούλιο, θα εργαστούμε αργότερα από ό,τι θα σα φαινόταν ε, κατάλληλο για να μην μείνουμε και πάλι ουραγοί. Ε, το Κοινοβούλιο να μπορέσει να πλαισιώσει μια φορά την εκτελεστική εξουσία και όχι αντιστρόφω. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι πολύ και θα είμαστε πραγματικά ε, πολύ πρόθυμοι να εξετάσουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώσαμε το σημείο 15. Να πάμε στο 25. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης για τους κανόνες αστικού δικαίου σχετικά με την ρομποτική. Ο λόγος στην εισηγητρία, την κυρία Ντελβού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τον Ιανουάριο του 2015 η Επιτροπή αυτή αποφάσισε να δημιουργήσει ομάδα εργασία για τις νομικές και δεοντολογικές συνέπειες της ρομποτικής. Είμαι ευτυχής που σήμερα μπορώ να σας αναφέρω το τι έχει συμβεί έκτοτε με το σχέδιο έκθεσής μου. Απεστάλλει χθε μόλις, με μια μορφή κάπως προσωρινή, ε, θα πρέπει να συμπληρωθεί από το αιτιολογικό σημείωμα, την αιτιολογική έκθεση, όμως ήθελα να τηρήσω το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει, να υποβληθεί τον Μάιο, γιατί εφόσον ξεκινήσουμε την ε, σχετική εργασία, φαίνεται ευθύ αμέσω ότι τα θέματα που άπτονται της ρομποτικής ξεπερνούν τις ε, καθεαυτές αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Οπότε θα σας αφήσω και χρόνο, συνάδελφοι, αλλά και στους συναδέλφους άλλων επιτροπών για να μπορέσετε να εξετάσετε το θέμα και να τοποθετηθείτε. Η προθεσμία ε, για την υποβολή τροπολογιών ορίστηκε τον Οκτώβριο, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας και πάνω απ' όλα τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής μας. Την νομική υπηρεσία, την υπηρεσία πολιτικών υποθέσεων και την ΣΤΟΑ η οποία εκπώνησε σχετική μελέτη για τις επιθυμητές και ανεπιθύμητες συνέπειες της ρομποτικής. Βλέπω την κυρία Βαν Βέντζελ που ε, μου υποσχέθηκε ότι η έκθεσή τους θα μας αποσταλεί σύντομα. Σε ό,τι αφορά το δικό μας το θέμα, διαπιστώνουμε ότι η αγορά της ρομποτικής αναπτύσσεται με ηλικιώδεις ρυθμούς και ότι όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια βιομηχανική επανάσταση. Κατά γενική γνώμη, ε, η ρομποτική είναι μια αγορά που θα έχει καθοριστική θέση σε όλες τις αγορές μελλοντικά και αυτό ήδη ισχύει σε πολλούς τομείς, τη δηλαδή μηχανική παραγωγή, τις μεταφορές, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη ήδη υπάρχουν, τα οχήματα χωρίς οδηγούς ήδη είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν στους δρόμους μας, βρίσκονται σε φάσεις ε, δοκιμασιών, αλλά και στη γεωργία, στις υπηρεσίες ε, προς τους πολίτες, την εκπαίδευση, για να μην μιλήσω για παιχνίδια, όπου τα ρομπότ είναι πανταχού παρόντα. Μιλώ έχοντας ε, διαγνώση. Τα ρομπότ λοιπόν θα γίνουν πιο ευφυή, πιο αυτόνομα και στο μέλλον. Δεν θα προγραμματίζονται για να παραλαμβάνουν πάντοτε την ίδια δράση, αλλά θα μαθαίνουν μόνο τους. Και θα λαμβάνουν και αποφάσεις θα επιδίδονται πια σε δραστηριότητες που ως τώρα αποκλειστικώς ε, προβλέπονταν και, και εκτελούνταν από ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια έχει καθυστερήσει στην παραγωγή των ε, βιομηχανικών ρομπότ και την παροχή υπηρεσιών. 32% της παγκόσμιας παραγωγής ρομπότ ε, το 2014. Βλέπουμε όμως ότι η Απονία, η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ισχυρότατοι ανταγωνιστέ. Εάν δεν θέλουμε η ευρωπαϊκή αγορά να κατακλειστεί από ρομπότ ξένης προέλευσης, από άλλες υπήρους και που δεν σέβονται τις δικές μας προδιαγραφές και τις αξίες μας, πρέπει η Ευρώπη να κινητοποιηθεί. Η πρόκληση για τον νομοθέτη είναι να παρακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις, το χαζόμενο στις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αρκετά ευέλικτο, ώστε να μην οδηγήσει σε ασφυξία τη βιομηχανία μας. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι και αρκετά αυστηρό ώστε να προστατευτεί ο καταναλωτή, αλλά όχι μόνο ο καταναλωτή. Οι πολίτε και η ανθρώπινη εξωπρέπεια καθώ και η κοινωνική μα συνοχή. Είναι θέματα που πρέπει να τα προσπιστούμε. Δεν θα μπω στι λεπτομέρειε τη κάθε μια πρόταση χωριστά, διότι χάρη στη συνεργασία όλων η έκθεση είναι σειρά αρκετά πλήρη, αλλά θα μπορούσε να πληρωθεί κι άλλο. Να σταθώ στα πιο ευαίσθητα σημεία. Μάλλον θα είναι αρκετά δύσκολο να εξασφαλίσουμε την προστασία του ιδιωτικού βίου. Η ροή ε, δεδομένων και η κατοχή δεδομένων. Τα ρομπότ δεν μπορούν να λειτουργήσουν εάν δεν είναι αλληλοσυνδεδεμένα. Έχουν ανάγκη από δεδομένα και εκεί θα πρέπει να υπαγρυπνούμε. Να επαγρυπνούμε να υπάρχει ισορροπία και ε, αναλογικότητα. Ε, θα πρέπει η αναλογικότητα να τηρηθεί για τη συλλογή και την τήρηση των δεδομένων. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η ασφάλεια. Δεν θέλω να αναλύσω και να μιλήσω εδώ για την ε, διαδικτυακή εγκληματικότητα, αλλά πρέπει να προσέχουμε ώστε τα ρομπότ από το σχεδιασμό τους και μόνοι και μόλις να συμπεριλαμβάνουν ε, μηχανισμούς προστασίας, ασφάλειας δηλαδή. Τυποποίηση λοιπόν θα χρειαστεί, αλλά και αποφυγή κατακαιρματισμού της ενιαίας αγοράς, της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Έχουμε βιομηχανικούς κλάδους, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, που είναι άκρος successful, έχουν μεγάλη επιτυχία, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η αγορά, η ενιαία αγορά μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα. Θα υπάρχει και το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, διότι ήδη υπάρχουν ρομπότ και θα δημιουργηθούν κι άλλα που μπορεί να παράγουν και έργα. Πώς θα ε, διευθυντήσουμε το θέμα αυτό του πνευματικού δημιουργού. Και επίσης το θέμα της υγείας. Τα ρομπότ μπορεί να καταλήγουν σε διάγνωση. Ποιος ήταν ο ρόλος των ιατρών. Μπορεί ε, ρομποτικές, ε, ρομποτικά μοσχεύματα να τοποθετούνται στους ανθρώπους μετά από ατύχημα. Το θέμα λοιπόν της υγείας και η όλη μας αντίληψη θα αλλάξει τελείως. Νομίζω ότι η δημιουργία κέντρων ρομποτικής σε όλα τα νοσοκομιακά ιδρύματα θα είναι κάτι που θα καταστεί αναγκαίο για να καλύψουμε αυτές τις μέρημνες. Η μεγάλη ανησυχία που επανέρχεται σε όλες τις συζητήσεις είναι αυτή της απασχόλησης, ωστόσο. Είναι πραγματικά μια μείζων ανησυχία, διότι τα ρομπότ μπορεί να κλέψουν τι θέσει εργασία των ανθρώπων. Οι ειδικοί είναι ε, διχασμένοι. 50% λένε ναι και 50% λένε ότι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση θα αντισταθμίσει την απώλεια των παλαιών. Δεν ξέρουμε καθόλου τι θα γίνει. Πώ θα συμφιλειώσουμε του ανθρώπου με τα ρομπότ, τι προσόντα θα χρειάζονται για να υπάρξει σωστή ενεργοδιάδραση. Και αν υποθέσουμε ότι και ε, κάποιε δύσει εργασία, σε τι θα εργαστούν αυτοί οι άνθρωποι, πώ θα απασχοληθούν, διότι η βιομηχανία τη ψυχαγωγία ε, μας δημιουργεί απορίες το πώς θα διοργανωθεί το μέλλον και για το πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Πρέπει να σκεφτούμε μια καθολική και πανανθρώπινη αμοιβή ενδεχομένως. Υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία που πρέπει να επιληθούν και είναι αρμοδιότητα τη δική μα επιτροπή. Είναι η ευθύνη που θα έχουν τα ρομπότ. Η σημερινή νομοθεσία δεν απαντά σε αυτό το είδο τις απαιτήσει που ε, προκαλούνται λόγω τη ρομποτική. Θα πρέπει λοιπόν στην Επιτροπή μα να υποβάλουμε μια πρόταση που να βασίζεται στην αυστηρή ευθύνη, ευθύνη που να ισχύει για τα ρομπότ ε, αυτή τη στιγμή, τα ρομπότ που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά και τα ρομπότ που θα ε, κατακλείσουν την αγορά τα ερχομένα χρόνια. Ε, έτσι, τίθεται και το θέμα της δημιουργίας και της υποχρεωτικής ασφάλειας για τα ρομπότ, όπως ε, συμβαίνει και με την ασφάλεια των αυτοκινήτων, και εάν δεν υπάρχει αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί και ένα ταμείο αποζημίωσης. Οι ασφαλιστικές, λοιπόν, θα ανθίσουν εδώ. Ταυτόχρονα η έκθεση ζητά να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, διότι νέα ρομπότ, όλο και πιο αυτόνομα, όλο πιο ανεξάρτητα και όλο πιο ευφυή, ήδη βρίσκονται στο στάδιο των πειραμάτων σε πολλά, εργαστήρια, σε πολλά ερευνητικά εργαστήρια στον κόσμο. Άρα θα πρέπει να αναλύσουμε ποιε θα είναι οι βέλτιστες λύσεις για να βρούμε απαντήσεις στα μελλοντικά προβλήματα. Θα πρέπει να έχουν προσωπικότητα τα ρομπότ με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε σήμερα. Αλλά θα πρέπει να το ε, έχουμε κατά νου. Δεν έχουμε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Όμως έχουμε την υποχρέωση να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην ε, παρακολουθήσουμε ως θεατές τους καταναλωτές να υπίστανται την εξάπλωση των ρομπότ σε όλους τους τομείς. Θα θέλαμε να είμαστε κάπως ε, πειθαρχημένοι στην προσέγγιση μας, δηλαδή να εντοπίσουμε τις διαφορετικές κατηγορίες ρομπότ για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε μητρώα και να τα καταγράφουμε, να τα ταυτίζουμε, να μπορούμε να τα ταυτοποιήσουμε. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας οργανισμός της ρομποτικής, ο οποίος να ε, τροφοδοτηθεί όχι μόνο με την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη στην τεχνολογία και τις επιστήμες, αλλά και την νομοθεσία και ενδεχομένως την κριτική. Ε, θα ήθελα επίσης να απευθύνω έκκληση προς την Επιτροπή και τα κρατημέλη που χρηματοδοτούν την έρευνα. Να μην γίνεται έρευνα μόνο για την τεχνολογία, αλλά να σκεφτούμε και τις κοινωνικές συνέπειες ε, με την έλευση όλων αυτών των ρομπότ. Όχι σε πέντε χρόνια, δεν θα γίνουν τότε αυτές οι αλλαγές. Ο ορίζοντας δεν είναι τόσο μακρινός. Σε 20-25 χρόνια θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Πρέπει λοιπόν να προετοιμάσουμε τις κοινωνίες μας σχετικά. Νομίζω ότι ρόλος μας είναι να ορίσουμε τις ε, θεμελιώδεις αρχές βάσει των οποίων θέλουμε να ε, αναπτυχθεί η ρομποτική. Εάν δράσουμε ταχαίως μπορεί να επηρεάσουμε μια διοργάνωση που θα ε, ισχύσει παγκοσμίω. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε να προσαρτηθεί και μια χάρτα με την σύσταση διοντολογικής επιτροπής και στα ερευνητικά κέντρα αλλά και για την θέση σε εμπορία και να δοθούν, να δίδει συμβουλές τους ε, χρήστες αλλά και τους παραγωγούς, τους κατασκευαστές των ρομπότ. Είναι σημαντικό λοιπόν να συμφωνήσουμε επί των αρχών αυτών και να παραμείνουμε σταθεροί στο μήνυμά μας και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προς την οποία απευθύνουμε έκκληση δράση, ανάληψης δράσης, αλλά και προς την βιομηχανία, η οποία πιστεύω ότι προσδοκά αυτούς τους ορισμούς μας και τις ε, πολιτικές μας συστάσεις. Διότι όλο περισσότερο αναπτύσσεται αυτός ο κλάδος, οπότε όλο και περισσότερο χρειάζεται και νομική ασφάλεια, ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο θα σταματήσω, θα πάυσω, ελπίζοντας ότι θα διαβάσετε με τα μεγάλη προσοχή στην έκθεσή μου και θα συμβάλλετε ε, με τις παρατηρήσεις σας ε, ώστε να γίνει πληρέστερη και πολύ πιο συγκεκριμένη. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεργαστούμε και θα μπορέσουμε όλοι μαζί να μελετήσουμε αυτό το θέμα. Ίσως μετά τις διακοπές. Ε, πρόεδρε, ολοκληρώνοντας να πω ότι η προθεσμία για την αποβολή των υπολογιών ορίστηκε στις 25 Οκτωβρίου ώστε να έχουν άφθονο χρόνο οι άλλες επιτροπές να συζητήσουν τη σχετική πρόταση και θα ήθελα η έγκριση στην Επιτροπή Γιούρη να προβλεφθεί για τις 29 Νοεμβρίου και να περάσει το θέμα στην Ολομέλεια στην τελευταία εβδομάδα του, του Δεκεμβρίου. Θα είναι ένα πολύ όμορφο χριστουγεννιάτικο δώρο. Ευχαριστούμε κυρία Κομοδίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω διατρέξει το σχέδιο της κυρίας Δελβό και νομίζω πραγματικά της αξίζουν ε, θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά της ως τώρα. Έχει ε, καλύψει πολλές από τις συζητήσεις που ήδη κάναμε στην ομάδα εργασία αυτή την και πολλές από τις συζητήσεις που έγιναν με πολλούς εμπειρογνώμονες επί του συγκεκριμένου θέματος. Νομίζω τα περισσότερα από όσα λέγονται, τα όσα δηλώνονται στην έκθεση αυτά, αυτή είναι μια γλαφυρή παρουσίαση και απήχηση των όσων ε, μας ε, συνέστησαν οι εμπειρογνώμονες και επίσης και των συζητήσεων που έγιναν σε αυτές τις ε, συνεδριάσεις. Μια πτυχή που ίσως και να χρειαστεί να της δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην έκθεση είναι οι συνέπειες της ε, εξέλιξης των ρομπότ και της αυξανόμενης χρήσης τους στην κοινωνική διάσταση του βίου μας, δηλαδή στον τρόπο ζωής μας, στο βιωτικό μας επίπεδο. Η έκθεση σωστά τονίζει τις δυσκολίες που θα προκύψουν στην απασχόληση. Επίσης, σωστά τονίζει και άλλες πτυχές όπου τα ρομπότ και η τεχνητή ευθεία θα προκαλέσουν αλλαγές ή τουλάχιστον έτσι αναμένεται. Θα έλεγα λοιπόν απλώς ότι προσωπικώς θα ήθελα να ε, τονιστεί και η κοινωνική διάσταση του βίου κάτι που πιστεύω ότι θα επηρεαστεί τα μάλα. Ε, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά γιατί υπάρχει πολύ σχετική προγνωμοσύνη και τεχνογνωσία. Όμως αυτά ε, ούτω ή άλλως θα είναι αντικείμενο και θύμα ανταγωνισμού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτόν τον ανταγωνισμό μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε μόνο να συνεχίσουμε να κρατομούμε και να αναπτύσσουμε τους δικούς μας τομείς. Οπότε, οπωσδήποτε πρέπει να παραμείνουμε στην επιπροστοφυλακή του σχετικού κλάδου και για να το πετύχουμε θα πρέπει όχι απλώς να εξεύρουμε κανόνες και να ε, δώσουμε στους ερευνητές και τη βιομηχανία μας ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο που σωστά εντόπισε και η συγκήτρια, αλλά Θέλω να πω, θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε για μια ισόρροπη προσέγγιση. Ισόρροπη προσέγγιση η οποία θα βοηθήσει όλους αυτούς να αναπτύξουν την ε, ρομποτική, να δημιουργούν, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε ότι οι ανθρώπινη αξιοπρέπεια και οι βασικές αρχές γίνονται σεβαστές. Νομίζω ότι η προτινόμενη έκθεση είναι ένα πολύ καλό σημείο αφετηρία για να αντιμετωπίσουμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίσουμε από τώρα τι μελλοντικέ προκλήσει. Όπω είπε και η συγκεντρία, υπάρχουν θέματα στα οποία δεν θα μπορέσουμε να βρούμε απάντηση τώρα. Σίγουρα και σήμερα, ενδεχομένω όχι και στο εγγύ μέλλον. Όμω, επειδή δεν είμαστε καν σίγουροι τι είδου αυτόνομα ρομπότ θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να την μεταστρέψουμε σε όπλο την αβεβαιότητα αυτή. Η δική μας δουλειά πρέπει να προβλέψει ένα ευέλικτο πλαίσιο. Ένα πλαίσιο τόσο διαλλακτικό που να μπορεί να προσαρμοστεί και να προσαρμόζεται στις διάφορες εξελίξεις ενώ λαμβάνουν χώρα. Θα κλείσω λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πλήρη, ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά για αυτόν τον κλάδο. Η ε, δυνατότητα διασύνδεσης για τα ρομπότ, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οχήματα χωρίς οδηγούς, πρέπει να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών, εάν θέλουμε πραγματικά να παραμείνουμε στην εμπροστοφυλακή αυτού του κλάδου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ, αλλά πρωτού δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδελφούς να σας θυμίσω ότι έχουμε λιγότερο από 30 λεπτά στη διάθεσή μας και έχουμε τουλάχιστον 4 ακόμη σημεία. Οπότε παρακαλώ, ο κύριος Άντερσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Τελβό είπε ότι ήταν χαρά της να παρουσιάσει την ε, έκθεση. Εμένα ήταν χαρά μου να το διαβάσω. Νομίζω ότι αντικατοπτρίζει πολύ καλά τη δουλειά που έγινε στην ομάδα εργασία. Είναι περίπου ένας χρόνος, και λίγο παραπάνω, που δουλεύουμε πάνω στο θέμα αυτό και από ό,τι φαίνεται τελικά φτάνουμε στο τέλος της αρχής αυτής της μακράς διαδικασίας. Νομίζω, πολύ σύντομα, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία της, ε, στην έκθεση που πάνε λίγο παραπέρα από ό,τι πρέπει. Το θέμα της ευθύνης, ας πούμε. Αν κάθε θέμα που ε, διαχειριζόμαστε το βλέπαμε με τον ίδιο τρόπο, η έκθεση αυτή δεν θα ήταν 19 σελίδες, θα ήταν 100. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει αρκετό περιθώριο να διευρύνουμε την έκθεση αυτή και να μπούμε σε περισσότερε πληροφορίε, λεπτομέρειε, συγγνώμη, για πολλά σημαντικά θέματα και νομίζω ότι είναι καλό που έχουμε χρόνο μέχρι την 5η Οκτωβρίου για να στείλουμε τις ε, προτάσεις μας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριο Καβαντά. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στάδιο αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση Κυρία Ντελβό, είναι εξαιρετική η δουλειά σας και η δική σας δουλειά και της ομάδας σας. Πραγματικά Έχετε συμπεριλάβει τα πάντα. Από την άλλη, αν πέρασε μία τόσο κακή συμφωνία, εσείς φταίτε. Οπότε και σας θαυμάζω, αλλά είμαι και λίγο εκνευρισμένος μαζί σας. Δεν είναι σαν τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε να εξετάσουμε. Είναι κάτι το οποίο είναι θεμελιώδου σημασίας ε, στο παρελθόν ε, ε, θα ήταν του, ε, της, της τάξεως ε, της ίδρυσης, της, της δημιουργίας των εμφολίων, της ανακάλυψης του ατόμου, της, του ηλεκτρισμού. Σε αυτή την κλάση θα, θα, θα έβαζα το θέμα της ρομποτικής. Με όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά και πολύ κακά πράγματα. Με το ατόμιο μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά μπορούμε και να σκοτώσουμε, ομοίως και με τα εμβόλια. Η ρομποτική λοιπόν είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους που εργάζονται σε τομείς που θα αντικαταστήσει η ρομποτική, ε, τι θα γίνει απλώς, θα γίνουν απλώς χειριστές των ρομπότ ή δούλοι των ρομπότ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Γιατί πάμε σιγά σιγά, αλλά δεν ξέρουμε πού είναι το όριο ε, υπάρχουν τεράστια πράγματα, τεράστια σημασία πράγματα που έχουν γραφτεί σε σχέση με, αυτήν, ε, την, ε, αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική ποιότητα και την προοπτική που έχετε συμπεριλάβει σε αυτή την έκθεση. Είναι πραγματικά καταπληκτική. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Στανμάιερ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκ μέρους της θα ήθελα να επικροτήσω την εξαιρετική πρωτοβουλία και τη δουλειά της ε, ομάδας του ΕΛΚ ε, υπό την ηγεσία της κυρίας Δελβό. Εμείς στο πλαίσιο της στρατηγικής είχαμε συμπεριλάβει, ότι, είχαμε πει ότι η αξιοπιστία στο πλαίσιο του διαδικτύου των αγαθών είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Ο στόχος της ψηφιακής αγοράς ε, της ε, ε, εσωτερικής, όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, είναι η προώθηση της ε, και ύπαρξη ενό σταθερού πλαισίου για, το, για, για τον κλάδο. Υπήρξαν πολλές διαβουλεύσεις το προηγούμενο φθινόπωρο μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους που αφορούσε πάρα πολύ το θέμα του διαδικτύου των ε, πραγμάτων και ε, του πλαισίου που πρέπει να υπάρχει, αλλά το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο καταλήξαμε ότι δεν είναι το κατάλληλο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των, ε, της, της ευθύνης του διαδικτύου των πραγμάτων. Ε, ανακοινώσαμε μία πρωτοβουλία ελεύθερης ροής πραγμάτων. Θα πούμε περισσότερα ε, κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πολλά σημεία όπως και το θέμα της ευθύνης ε, και άλλα θέματα όπως η κυριότητα των δεδομένων και συμβάσεις μεταξύ μηχανών κλπ. Επίσης θα τονιστούν σε αυτήν την έκθεση που θα υποβάλουμε. Έχουμε ήδη προβεί σε, κάποια, σε κάποιες πρωτοβουλίες 80 εκατομμύρια διατίθενται σε ερευνητικά προγράμματα από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ' έτος. Έχουμε ένα πάρα πολύ περιεκτικό χαρτοφυλάτιο που καλύπτει τα ιατρικά ρομπότ, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη κλπ. κλπ. Όλα αναφέρονται σε αυτή την έκθεση. Και επίση για τα αυτόνομα ε, οχήματα προσπαθούμε να, να δούμε πώς θα γίνουν δραστηριότητες πολλαπλών ελέγχων. Ε, σε σχέση με όλα αυτά που ανέφερε η κυρία Ντελβό, θα ε, εγκριθεί σχετικός κανονισμός και φυσικά θα υπάρξει περαιτέρω προστασία προσωπικών δεδομένων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ε, πραγματικά ατενίζουμε μαζί με σας το μέλλον της συνεργασίας μας για το θέμα αυτό. Ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης αλλά και από την Γενική Διεύθυνση Connect θα ε, εξετάσουμε από κοινού όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι ευρύτατα, όπως είπε και η κυρία Ντελβό, για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες λεπτομερείς συζητήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος και εγώ ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Οπότε δεν ξέρω, κυρία Ντελβό, θέλει κάτι να πει. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, το καταλαβαίνω, οπότε θα ήθελα να επαναλάβω ε, ότι ε, με χαρά θα ολοκληρώσω την έκθεσή μου, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία που άκουσα. Περνάμε τότε στο σημείο 27 της τη διάταξης, λέει ο Πρόεδρος. Ερμηνεία και υλοποίηση της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Εγώ πρέπει να το κάνω αυτό. Σύντομο θα είμαι, όπω γνωρίζετε, στι 13 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, υπέγραψαν ε, διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας και η δική μας Επιτροπή και Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων αποφάσισε να ιδρύσει μια κοινή ομάδα εργασίας για την ερμηνεία και την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας όπως επίσης και με σκοπό την προετοιμασία μιας έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας για το ίδιο θέμα Υπάρχουν δύο συνεισηγητές, ε, ο κύριος Κόρμπετ εκ μέρους της Επιτροπής ΑΦΚΟ και ο υποφαινόμενος εκ μέρους της δικής μας Επιτροπής. Στις 10 Μαΐου του 2016 η ομάδα εργασίας ε, είχε την πρώτη της ε, συστατική επιτροπή όπου ενέκρινε την ε, δήλωση αποστολής της και ε, με κατανόηση βέβαια του γεγονότος ότι και τα δύο αυτά έγγραφα είναι ζωντανά, τα οποία θα ενημερώνονται ε, βεβαίως σύν το χρόνο αν χρειαστεί. Στην πρώτη μας αυτή συνεδρίαση, λοιπόν, ακούσαμε την παρέμβαση της κυρίας Φραντσέσκα Ράτη υφυπουργό ε, της μάλλον, συγγνώμη, αναπληρωτή, ε, Ανατεπιληρώτρια ε, διευθύντρια ε, του οργάνου ελέγχου της διοργανικής ε, συμφωνίας και ελπίζουμε ότι η επόμενα συνεδρίαση θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο. Να σας ενημερώσω επίσης ότι εντωμεταξύ η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να ιδρύσει μία ακόμη ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό. Αποφάσισε λοιπόν να ορίσει τους προέδρους της ε, Γιούρη και, τους, και της Ράφκο, δηλαδή α, και τους δύο συνεισυχητές, ε, ε, τον κύριο Κόρμπετ και τον κύριο Φερχόφστατ, ως μέλη αυτής της νέας ομάδας εργασίας. Και εμείς έχουμε προσκληθεί στην επόμενη διάσκεψη των Προέδρων για να, για να ε, διευθετήσουμε τις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε με την επιστολή του κυρίου Μπούζεκ εκ μέρους του CCC, ο κύριος Σάρε, ε, Σάρε να είναι ο υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση της, του ορισμού των κριτηρίων, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν ε, με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων της Γιούρη και όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες, επίσης να, να ακολουθήσουμε ε, το CCC ώστε οι επιτροπές ίντα ε, και ΑΦΕΤ, μάλλον οι πρόεδροι των επιτροπών αυτών, να ε, πρωτοστατήσουν στις διαπραγματεύσεις. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ σε σχέση με την ε, υποβολή έκθεσης που έπρεπε να σας κάνω για το θέμα αυτό. Μήπως υπάρχουν ιδέες, διαφωνίες, παρατηρήσεις. Όχι. Πολύ ωραία. Προχωρούμε άρα στο σημείο 28. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την επίτευξη του ορίου για την κίνηση της διαδικασίας κίτρινης κάρτας όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Δίνω το λόγο στον κύριο Λεμπρετών που είναι ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είναι ένα κείμενο πάρα πολύ σημαντικό ε, το οποίο εξετάζουμε εδώ γιατί αφορά ένα σχέδιο τροποποίησης ε, της ε, περιβόητης οδηγίας του 2016 για την απόσμαση εργαζομένων. Νομική βάση είναι η ίδια με αυτήν, για την οδηγία αυτή, 53, το άρθρο 53 δηλαδή από το, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν πω σε λεπτομέρειες τεχνικές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τονίσω εισαγωγικά ότι από πολιτική απόψεω εγώ διαφωνώ με αυτήν την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων και συνεπώ διαφωνώ και με την τροποποίησή τη. Αυτή η τροποποίηση σκοπό έχει να υπάρξουν κάποιες διευκρινήσεις, σας υπενθυμίζω τις βασικές, το δικαίωμα εργασίας, ε, του τόπου εργασίας θα ισχύει για τους αποσπασμένους, ε, τα ίδια θα ισχύουν δηλαδή και για αυτούς τους εργαζόμενους. Ε, οι μισθοί τους πρέπει να είναι οι ίδιοι με τους μισθούς των ε, ντόπιων εργαζομένων. Ε, πρέπει επίσης να τα λάβουμε υπόψη κατά την, τον καθορισμό των μισθών τους και επίσης έχει να κάνει αυτό και με την η υπεργολαβία και τη δυνατότητα προσφυγής σε διασυνοριακό επίπεδο. Ε, υπήρξαν αιτιολογημένες γνώμες ε, από 11 ε, κράτη-μέλη, οπότε περνάμε το κατώτατο όριο. Δανία και ανατολικές χώρες έστειλαν αιτιολογημένες γνώμες, γιατί αυτή είναι, είναι υπάροχοι υπηρεσιών και θεωρούν ότι ε, με την τροποποίηση θίγονται όλος ιδιαίτερος γιατί θα μειώσει, τέλος πάντων υπάρχει ο κίνδυνος μείωσης του αριθμού των αποσπασμένων εργαζομένων. Τα επιχειρήματα που ε, παρατίθενται είναι πολλά, δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα, όμως είναι, είναι ενδιαφέροντα και γι' αυτό θα ήθελα να τα ομαδοποιήσω σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον, μία, εν υπάρχει ένα επιχείρημα διαδικαστικής φύσεως που συνδέεται με το γεγονός ότι σύμφωνα με πολλά από αυτά τα κράτη-μέλη είναι πρόημη αυτή η τροποποίηση, γιατί κατά τη γνώμη τους θα έπρεπε να περιμένουν να ολοκληρωθεί η περίοδος μετάβασης προηγούμενης οδηγίας για να περάσουμε στην επόμενη. Όμως αυτή η προηγούμενη οδηγία είναι αυτή του 2014, εκτελεστική ε, του, για το 2016 και εκπνέει στις 18 Ιουνίου του 2016. Να λοιπόν ένα ενδιαφέρον νομικό επιχείρημα, ένα πρώτο ενδιαφέρον νομικό επιχείρημα, δεν ξέρω ποια είναι η άποψη της ε, Επιτροπής, ε, εγώ προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ πεπισμένος, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να εξετάσουμε, μπορούμε να εξετάσουμε παράλληλα αυτήν την τροποποίηση, παρά το γεγονός ότι δεν έχει περάσει ακόμη η ε, προθεσμία, η μεταβατική της προηγούμενης. Δεν μας εμποδίζει κανείς να κάνουμε την εξέταση αυτή. Επόμενη ομάδα επιχειρημάτων, η επικουρικότητα τέσσερα επιχειρήματα τα οποία μου φαίνονται ενδιαφέροντα και ε, σχετικά και δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Πρώτο επιχείρημα η αμοιβή των εργαζομένων ε, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και αυτό ε, το λέει η Δανία, αυτό είναι το επιχείρημα της Δανίας που διαπιστώνει και αυτό είναι ενδιαφέρον ότι η φράση που εξασφάλιζε ότι πολιτική εθνική είναι η αμοιβή των εργαζομένων έχει απαλληφθεί από το κείμενο. Εδώ λοιπόν υπάρχει ε, μία επιπλέον ε, διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Δεύτερο επιχείρημα είναι η έννοια του ίσου, ε, της ίσης αμοιβής, ε, κάτι το οποίο μειώνει την ελεύθερη ε, κυκλοφορία των ανθρώπων και των υπηρεσιών, κάτι το οποίο ανέφερε η Εστονία. Τρίτο επιχείρημα, η έννοια της αμοιβή που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό είναι αμφίσιμη σε αντίθεση με την προηγούμενη έννοια του ελάχιστου του, του μισθού. Ε, αυτό είναι νομικής φύσεως, ε, βέβαια, είναι αυτό το οποίο ε, λέει η Ουγγαρία και λέει μάλιστα ότι αντιβαίνει στην επικουρικότητα. Τέταρτο επιχείρημα, που είναι και το πιο ευνόητο, το πιο εύληπτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατηγορείται ότι ε, παρεμβαίνει ε, σε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών ε, ε, και η Τσεχία το, το παρέθεσε αυτό το επιχείρημα και αυτό εξηγεί και για ποιο λόγο ξεκίνησε η διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Έτερα επιχείρημα ε, αφορά την αναλογικότητα, λιγότερο σημαντικά είναι αυτά, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό και ενδιαφέρον από τη Λετωνία που λέει ότι είναι δυσανάλογο να περνάμε από την απλή υποχρέωση ενός ελάχιστου μισθού σε μία πιο απαιτητική αρχή ίσης αμοιβή για τους αποσπασμένους ε, εργαζομένους. Εδώ λοιπόν γίνεται λόγος δυσανάλογης προσέγγισης ε, για να επιτύχουμε έναν στόχο. Ε, υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες ε, συμφωνούν σε αδρές γραμμές με τη Λετωνία χωρίς να το θέτουν τόσο καλά το επιχείρημα αυτό ότι δεν είναι δυνατόν με, κάποιο κανονισμό, με κάποια τροποποίηση νομοθετικής πράξης να ορίζεται ο μισθός των ανθρώπων, γιατί εκεί ε, αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι έρχεται να παρέμβει στην, ε, στον ελεύθερο ανταγωνισμό και στην ε, ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Ε, επίσης, τα κοινωνικά, οι κοινωνικές εισφορές ε, εξακολουθούν όμως να πληρώνονται στη χώρα ε, προέλευσης των αποσπασθέντων εργαζομένων, κάτι που σημαίνει ότι είναι σε πλεονεκτική σχέση με, σε σχέση με τους ντόπιου εργαζόμενους ή αποσπασμένοι. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα επιχειρήματα και πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Σλοτόφσκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή τη διεξοδική παρουσίαση. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια επιχειρήματα από την πλευρά της Πολωνίας. Όπως θα ξέρετε, η Ένωση δεν αποτελείται από κράτη-μέλη που έχουν το ίδιο επίπεδο ΑΕΠ ή μισθών. Είναι προφανές και πρέπει να το γνωρίζουμε ενώ συζητούμε τις προτινόμενες τροπολογίες για την οδηγία. Βεβαίως θα ήταν απλούστερο να κάνουμε σχέδια για το κοινό μας μέλλον, να ήταν διαφορετική κατάσταση. Όμως έτσι έχουν τα πράγματα, τι να κάνουμε. Και τα παλαιά και τα νέα κρατημέλη το γνώριζαν ανέκαθεν. Ναι, Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας και τις αποκλήσεις μας, αλλά όσο περισσότερο προσεγγίζουμε τα κοινά μας ιδεώδη, όλο τόσο περισσότερα εμπόδια ξεπηδάνε. Βλέπουμε να υπάρχει τάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα αποτελεί διάκριση Βεβαίω καταλαβαίνουμε ότι έχει καλέ προθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ταυτόχρονα φοβούμεθα ότι υπάρχουν παλιά ένστικτα προστατευτισμού που αναβιώνουν εδώ. Θα πρέπει η διαδικασία τη κίτρινη κάρτας να κάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί εάν θέλει να ανταγωνιστεί κατά αυτόν τον τρόπο τα κράτη-μέλη ή όχι. Η Πολωνία είναι ηγέτη στον τομέα των ε, ε, υπηρεσιών που παρέχονται από τους ε, εργαζομένους. Θέλουμε λοιπόν καλή ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους εργαζομένους επίσης, είτε είναι Εστονοί, είτε Πολωνοί, είτε Τσέχοι. Και επίσης πολλοί έρχονται στην περιοχή μας, όχι μόνο λόγω του χαμηλότερου κόστους, και για τους δικούς τους λόγους, αλλά δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε. Γι' αυτό έτσι λειτουργεί η εσωτερική αγορά. Είμαι κατά της ιδέας να αφαιρέσουμε δικαιώματα των δικών μας εργαζομένων να ανατρέχουν σε αυτό το μηχανισμό. Έχουμε την παλιά οδηγία για την προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων κατά των ε, μορφών διακριτική μεταχείρισης και εφόσον ισχύει πρέπει να πούμε ότι προτείνει κάτι καινούριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κατά της επικουρικότητα. Έχουμε δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αγνοεί την αρχή της επικουρικότητας ε, παρελειμμένως. Σε αυτή την περίπτωση Το γεγονός ότι έχουμε κάνει αυτή την πρόταση σημαίνει ότι μπορούμε να παρεμποδίσουμε τέτοιες ατασταλίες. Θέλω λοιπόν να καλέσω όλους να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Πρέπει να προτεύσουμε και τις αγορές μας. Πριν δώσουμε το λόγο στους επόμενους ομιλητές, πρέπει να αναβάλουμε τα επόμενα δύο σημεία που έχουμε στην εμερήσια διάταξη, μετά από το, τότε σημείο λοιπόν. Πάμε στον κύριο Νίλσον πρώτα. Έξι λεπτά έχουμε παρακαλώ. Βεβαίως πολύ σύντομα πρόεδρε. Συνήθως ε, ε, δουλεύω στην τρένο που ήμουν υπεύθυνο για την γνωμοδότηση για το κοινωνικό ντάμπινγκ, για, την, ε, για τις αποσπάσεις των εργαζομένων. Το θέμα αυτό είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητο και πολύ περίπλοκο. Γιατί υπάρχουν πολύ ευρείε απόψει. Αυτό που δείχνει η κίτρινη κάρτα είναι ότι υπάρχουν ισχυρές απόψεις για το θέμα αυτό και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ενώ τα εθνικά κοινοβούλια που εκδίδουν την κίτρινη κάρτα έχουν ε, θίξει πολύ σημαντικά θέματα όπως η ελευθερία της μετακίνησης, ε, η ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών, αυτό δεν είναι θέμα επικουρικότητας. Η πρόταση ασχολείται με ήδη υπάρχουσα νομοθεσία, κείμενη νομοθεσία που αποδείχθη αρκετά προβληματική για κάποιε χώρε και από τη δική μου την πλευρά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ίσω ίση μισθοδοσία για την ίδια δουλειά. Η πρώτη κομισιόν πηγαίνει προ σωστή κατεύθυνση και πρέπει να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. Η έκθεση, της, ε, η έκθεση Λαβάλ και ο ε, της ε, φάνηκε ότι επηρεάζει τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις συλλογικές ε, διαπραγματεύσεις, ε, κυρίως για, την, ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θέμα αυτό δεν μπορούμε να, το, να μην το διαχειριστούμε επειδή είναι απλώς ευαίσθητο, αλλά πρέπει να βρούμε ένα συμβασμό ο οποίος το δουλεύει για όλους. Θέλω λοιπόν να ενθαρρύνω την Κομισιόν να μην αποσύρει την πρότασή της, ούτε να την αποδυναμώσει, την έχουμε συζητήσει και πρέπει να τη συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ, περιοριστείτε σε ένα λεπτό. Η κυρία Ρέγνερ. Δύσκολα, Πρόεδρε, θα περιοριστώ σε ένα λεπτό για αυτό το θέμα. Γιατί έχουμε αυτή την πρόταση. Επειδή προέκυψαν καταπατήσεις και επειδή μιλούμε για την ελεύθερη μετακίνηση. Μία από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες που μας ε, κάνει να ζητούμε μια συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα αυτό, κυρίω για διασυνοριακέ αποσπάσει. Ή όλο και περισσότερε χώρε εμπλέκονται σε κάτι τέτοιο. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι γίνεται σε μια χώρα, αλλά σε πολλέ χώρε συμβαίνει αυτό. Και πάντα το θέμα είναι η αναλογικότητα και η επικουρικότητα που πρέπει να εξετάζονται. Γιατί ακριβώ εδώ μιλούμε για αδυναμία διαχείριση του συστήματο χωρί να έχουμε μια ευρωπαϊκή ε, ρήτρα γι' αυτό. Τώρα, να σα θυμίσω ότι υπάρχει θεμητό ανταγωνισμό, υπάρχει και αθέμητο ανταγωνισμό. Και ο στόχος ε, είναι ακριβώς να αποφύγουμε το ε, ε, κοινωνικό ντάμπινγκ, το ντάμπινγκ των μισθών. Να μπορέσουμε να το προλάβουμε επίσης. Και γι' αυτό Αυτό γίνεται στα πλαίσια της, των συνήθων αρμοδιότητων της ε, Κομισιόν και βεβαίω τα στοιχεία αυτά στην πρότασή της θα πρέπει να ενισχυθούν. Ευχαριστώ η κυρία Γκέφχαρτ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όντως εδώ πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να έχουμε κάτι ως δεδομένο. Ο στόχος αυτής της οδηγίας είναι να απαντήσει στην κινητικότητα και στη διασυνοριακή εργασία. Αυτά, περσέ, είναι θέματα που δεν μπορούν να τύχουν εθνικής διαχείρισης αλλά πρέπει να τα, να τα διαχειριστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως είπε και η κυρία Ρέγνερ και έχει δίκιο, πρέπει να αποφύγουμε να υπάρχουν ε, καταπατήσεις των δικαιωμάτων των ε, πολιτών και βεβαίως υπάρχει και η οδηγία για τις υπηρεσίες και, αυτός, και αυτές οι δύο συζητήσεις συνδυάζονται γιατί πρέπει βεβαίως να αποφύγουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των κοινωνικών συστημάτων των κρατών μελών. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, αυτό ακριβώς, και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Άλλο ένα σημείο είναι ότι υπάρχουν νέα ε, επιχειρησιακά μοντέλα με αυξανόμενες τάσει, κυρίω στα πλαίσια αυτής της ψηφιακή δυνατότητας που υπάρχει για διασυνοριακή εργασία και επίσης και αυτό θα πρέπει να το δούμε και να το εντάξουμε στη συζήτησή μας. Και βεβαίω το θέμα της ε, επικουρικότητα είναι ότι εδώ ακριβώς πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση. Βεβαίω υπάρχουν λαϊκιστικέ απόψει στην ε, Ευρώπη και σε αυτέ θα πρέπει να στείλουμε μια σαφή απάντηση έτσι ώστε να πιστέψουν και οι πολίτε ότι πρέπει όντω να υπάρξει καλύτερο κοινωνικό μοντέλο. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το προωθήσουμε ενεργά. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σαϊέρ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα να επικεντρωθώ στο εξή. Έχω τι απόψει μου εγώ για το θέμα αυτό και βεβαίω ε, κατανοώ την μπορεί να επιστρέψει πίσω στην Επιτροπή η συζήτηση και να, για να δούμε και κάποια κοινωνικά θέματα. Συμφωνώ με του συναδέλφου που λένε ότι η πρόταση αυτή αντίκειται στι αρχέ τη αναγκαιότητα και τη ε, αναλογικότητα και θα περιορίσει την ελευθερία να παρέχονται υπηρεσίε, θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό κλπ. Αλλά επειδή είμαστε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις νομικές πτυχές αυτού του θέματος. Οι άλλες ε, επιτροπές βεβαίως έχουν εμπειρογνωμοσύνη στις υπόλοιπες ε, διαστάσεις του θέματος. Επίσης, άλλο ένα θέμα είναι ότι πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την διαδικασία της κίτρινης κάρτας, η οποία είναι ένα ζήτημα σημαντικό νομικής υφής. Έχουμε μια πρόταση εδώ η οποία ρυθμίζει θέματα που ήδη ρυθμίζονται ειδικά από τον κανονισμό Ρώμη 1, ελευθερία επιλογής ε, ενοχικού δικαίου. Ρώμη 1, 3 και 8 άρθρα. Που είναι ουσιαστικά νομικό θέμα που πρέπει να το απαντήσουμε. Είναι μια οδηγία αυτή που θέλει να ρυθμίσει πράγματα που ήδη ρυθμίζονται από τον κανονισμό. Και μπορεί να προκύψει νομική αβεβαιότητα. Άλλο ένα θέμα. Το θέμα της αποζημίωσης αντί για ε, ε, ε, επιχρήμαση. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα. Η αποζημίωση είναι όρος που ορίζεται αλλά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει αβεβαιότητα. Οπότε εμεί νομίζω ότι καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε και την νομική υπηρεσία και ω Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι κάποιε από αυτέ τις νομικέ πτυχέ. Και έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την απόφαση του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να το συζητήσει το θέμα αυτό, αλλά έτσι νομίζω πως πρέπει να πράξουμε εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα για το θέμα αυτό. Ε, υπάρχει παραβίαση της αρχής επικουρικότητας και αναλογικότητας από τη μία και από την άλλη η οδηγία αυτή περιλαμβάνει πολλά προβλήματα γιατί παραβιάζει και την συνθήκη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο υπογράμισε υπογραμμίστηκε σε σχετική έκθεση της ε, ε, Ρουμανίας. Ε, η Ρουμανία επηρεάζεται πολύ από την οδηγία τούτη και υπάρχουν πολλά προβλήματα που προκύπτουν από αυτή την οδηγία γιατί επηρεάζει τις διαδικασίες απόσπασης εργαζομένων, δημιουργεί προσκόμματα, τύχη στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Πρέπει να είναι σαφή τα πράγματα. Ο αριθμός των συμβάσεων, αν περάσει οδηγία, θα μειωθεί. Και άρα θα μειωθούν και οι θέσεις εργασίας, που προφανώς αντίκειται στο σχέδιο Juncker. Τέλος, η αρχή αυτή της ε, ίσης, ε, του ίσου μισθού για την ίση ε, δεν συνάδει με την ενιαία αγορά, γιατί οι διαφορές στους μισθούς είναι θεμητό στοιχείο του συγκριτικού πλεονεκτήματος των παρόχων υπηρεσία. Ευχαριστώ. Mr. Zwiefka. Ο κύριος Βιέφκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο θέματα. Καταρχάς υποστηρίζω πλήρως τον κύριο Σέγερ. Όντω, το θέμα αυτό ορίζεται, ε, συνδέεται με, τον, με την αλλαγή στον ορισμό στο άρθρο 2. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Η πρόταση τη θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Τώρα, αν μιλούμε για τη Ρώμη 1, πώς φαντάζεστε ότι η οδηγία μπορεί να αντικαταστήσει έναν κανονισμό. Είναι παράλογο και νομίζω ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να το ξέρουν. Γιατί αγνοείτε τη, νομική, αγνοείτε δική σας νομική υπηρεσία η οποία ε, τα, ε, τάχθη αναφανδόν αντίθετα με αυτό που παρουσιάσατε. Και συμφωνεί με αυτούς που λένε ότι η οδηγία δεν μπορεί να αλλάξει τις διατάξεις που περιλαμβάνει ο κανονισμός. Κανονισμός που είναι ενισχύει στα κράτη-μέλη. Εμπαρόδο. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου να προετοιμάσει μια γνωμοδότηση επί του θέματος αυτού, γιατί γνωρίζουμε ότι η γνωμοδότηση της, Ευρωπαϊκής, ε, της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρνητική. Είναι καλό λοιπόν που κάνουμε την ανταλλαγή απόψεων σήμερα, αλλά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε δουλειά πάνω σε τούτη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται από τη συνθήκη να παρουσιάσει μία επίσημη θέση. Ακριβώς ε, λόγω της εκκρεμούσας διαδικασίας της κίτρινης κάρτας. Η Κομισιόν μπορεί να αποσύρει την πρότασή της, μπορεί να αλλάξει την πρότασή της, να την τροποποιήσει ή μπορεί να την διατηρήσει, να διατηρήσει την παρούσα κατάσταση και να αποφασίσει ότι είναι σοφότερη από οποιονδήποτε άλλον. Αλλά αυτό θα πρέπει να ε, δηλωθεί επισήμω και δημοσίω. Πριν γίνει κάτι τέτοιο, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα ζητήσουμε τη γνώμη του, της υπηρεσία, όπω όπως είπατε. Πριν δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λεμπρέτο, να πω δύο πράγματα. Θα πρέπει να δούμε λίγο τη γενικότερη εικόνα για τούτη την πρόταση. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει ο ίδιος μισθός για, το, για την ίδια θέση εργασίας. Ε, αν θέλουμε θεμητό ανταγωνισμό, γιατί δεν έχουμε ίδιο μισθό για την ίδια θέση εντός της ίδιας εταιρεία. Μία πτυχή του θέματος είναι αυτή. δεύτερη πτυχή. Η αρχή αυτή είναι καλή Εφόσον όμως ε, δούμε τις, ε, τις διαπραγματεύσεις με, την, ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο και τα ωφέλη εντός της εργασίας, πολλές φορές βλέπουμε εντελώς αντίθετα πράγματα να συμβαίνουν σε σχέση με τότε την αρχή που συζητούμε. Δύο πολύ σύντομα σχόλια από δικιά μου πλευράς και να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Λεμπρετό. Oui, une conclusion très brève. Ναι, ένα πολύ σύντομο συμπερασμά. Η συζήτηση μόλι επιβεβαίωσε αυτό που είχα αρχίσει και εγώ να λέω με έμφαση. Ε, ελπίζω να το επιβεβαιώσει και η νομική υπηρεσία. Διαρωτώ με αν μια λύση για να προχωρήσει το όλο θέμα δεν είναι να αποφύγουμε. Να επουσκαλέσουμε, συγγνώμη, τον αρμόδιο επίτροπο στην επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Πολύ καλή ιδέα. Η συζήτηση αυτή πρέπει να συνεχιστεί σε μια από τι επόμενε συνεδριάσει. Πρωτού ολοκληρώσουμε την σημερινή συνεδρίαση, να σα ενημερώσω. Τα σημεία 36 και 37 δεν έχουν καμία αντίρρηση που να τα βαραίνει, όπως μας είπε η κυρία Κάουφμαν που δεν είναι εδώ, οπότε δεν χρειάζεται καν να τα συζητήσουμε Μόνο τα σημεία του κυρίου Λεμπρετού αναβάλλονται μέχρι την επόμενη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσελευσή σας και θα συναντηθούμε και το απόγευμα στην κοινή συνεδρίαση με την ΙΜΚΟ.